Λοιπόν, σα καλωσορίζω και πάλι όλου και σα καλημερίζω. Σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, ήθελα να θυμίσω ότι έχει γίνει μια αλλαγή. Χτες, δεν είχαμε την έκθεση ε, ε, τη δυνατότητα μάλλον να διεκπέρασουμε την έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου για την Όλαφ. Θα το κάνουμε σήμερα στις 2.30 το απόγευμα για να μπορέσει να μας ενημερώσει ο κύριος Μαρινέσκου ε, σχετικά με τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που είχε για την Όλαφ. Και θα περάσουμε στο σημείο 9 στην, της ημερήσιας διάταξης. Θα ακούσουμε τον Άλεξ Μπρένικ Μέιερ που είναι υποψήφιο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως γνωρίζετε ανανεώνεται μερικώς η σύνθεση. Η συγητής μας είναι ο κύριος Στεχόφσκι. Α, έχει έρθει ο υποψήφιος ήδη και κάθε δίπλα μου, δεν σας είδα. Σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Μπρένιγκ Μάιερ λοιπόν θα πάρει πρώτο το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Χόλμαια και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας συστηθώ ως υποψήφιος για μια δεύτερη θητεία ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θέλω να συστηθώ στην Επιτροπή σας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, Πρώτον, έχω πλήρη ευθύνη ε, των πεπραγμένων μου ως μέλος την τελευταία εξαετία και δεύτερον θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα τα κίνητρά μου και τις προθέσεις μου για το επόμενο διάστημα. Πριν από έξι χρόνια που είχα ξαναέρθει στην Επιτροπή σας, όπως και σήμερα, είχα κάνει δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, παρατήρησα ότι οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου ήταν ασαφείς ακόμα και αν κάποιος ε, που ενδιαφέρεται πολύ αλλά δεν είναι εντός ε, ε, των πραγμάτων έχει μεγάλες δυσκολίες να καταλάβει την ουσία των μηνυμάτων. Ως μέλος ανέκαθεν δραστήρια ήμουν υπέρμαχος μιας απλής γλώσσας για τις ετήσιες εκθέσεις μας και τις ειδικέ εκθέσεις. Έχουμε μια σύντομη έκθεση εκλεκευμένη που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο και αυτό δείχνει πόσο θετικά αποτελέσματα είχαν οι προσπάθειε μου καθώς επίσης και του ίδιου του ελεκτικού συνεδρίου. Και πάλι πριν από έξι χρόνια η δεύτερη μου παρατήρηση ήταν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, το ελεκτικό συνέδριο επί 20 χρόνια εξέδιδε αρνητική ε, γνωμοδότηση για τα ευρωπαϊκά ε, οικονομικά. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια έπαιρνε απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κάπως μπέρδευε τον έξω κόσμο με την ε, αναθεώρηση ε, της δήλωσης αξιοπιστίας τα τελευταία χρόνια το μήνυμα έχει γίνει πια πιο ρεαλιστικό και η ενημέρωση του συνεδρίου προς το Κοινοβούλιο ως προς τις αδυναμίες, ε, ε, τα νομικά ζητήματα και τις παρατυπίες στην διαχείριση των οικονομικών έχει βελτιωθεί σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, η σαφήνεια στη γλώσσα και η αναθεώρηση της δήλωσης αξιοπιστίας ε, είναι κομβικά για τη στρατηγική μας 2018-2020. Προείδρευσα στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας και ήμουν και εισηγητής. βασική στόχη της ε, λόγω στρατηγικής είναι να ε, δαπανώνται λιγότεροι πόροι για την, τις εκθέσεις για τη συμμόρφωση και περισσότεροι για τις εκθέσεις πεπραγμένων και επιδόσεων. Και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μα με τον έξω κόσμο, ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Η λογιστική έκθεση για την απλούστευση του ορίζοντα 2020, για την οποία ήμουν εισήγητή, καταδεικνύει τη σημασία της νέας αυτής στρατηγική. Κάθε χρόνο το ε, ελεκτικό συνέδριο δήλωνε ότι ο δείκτης φαλμάτων για τον ορίζοντα 2020 ήταν ανάμεσα στο 4 και 5%. Και κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο εξέφραζε την ενόχλησή του ε, για αυτό τον υψηλό δείκτη σφαλμάτων. Ω εισηγητή για το κεφάλαιο αυτό στην ετήσια έκθεση, ανέλησα για ποιο λόγο ήταν τόσο υψηλό αυτό ο δείκτη σφάλματο και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ε, βασική αιτία ήταν οι περίπλοκοι κανόνες για την έγκριση της χρηματοδότησης. Γι' αυτό άρχισα να ε, προτείνω την ε, απλούστευση για τον ορίζοντα 2020 και το ορίζον Ευρώπη στη συνέχεια. Έκανε συστάσεις στο Ελεκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ενέκρινε ως πολύ χρήσιμες γιατί συμπεριλήφθησαν στην νομοθετική διαδικασία. Ωστόσο, η μετάβαση της δήλωσης αξιοπιστίας μας ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Μία από τις φιλοδοξίες μου για τα επόμενα έτη είναι να συνεισφέρω έτσι ώστε ε, να γίνει πιο λογική η μεθοδολογία μας για τη δήλωση αξιοπιστίας. Ετησίως δαπανούμε πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ ε, για την εκπόνηση της δήλωσης αξιοπιστίας. Αυτό το ποσό είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μου, 60 εκατομμύρια, δεδομένου ότι είναι περιορισμένες οι πληροφορίες μας ε, στην ετήσια έκθεση και εξίσου συνεπώς περιορισμένη και η επίδραση και ο αντίκτυπο. Επίση, είμαι μέλο τη ψηφιακή επιτροπή που εργάζεται για την ψηφιοποίηση ε, τη δήλωση αξιοπιστία μα. Επιπλέον, πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε συστηματικά τη μεθοδολογία μας και ε, να αποφύγουμε μονομερή αναζήτηση σφαλμάτων οι εκθέσεις μας θα πρέπει να είναι ενημερωτικές και κριτικές, ε, ε, αλλά πάντα ισορροπημένες. Αν με ρωτάτε ποια είναι τα κίνητρα μου, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο δημοκρατικό έλεγχο που ασκεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εγκαίρως να ενημερώνεται σωστά για του λογαριασμούς και τις επιδόσεις των διαφόρων προγραμμάτων πολιτικής. Για το λόγο αυτό, η καλή επικοινωνία με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δικαιούχους ε, στα κράτη-μέλη είναι εκ των ουκάνευ. Για τα τελευταία έτη είχα την πρόθεση να υπηρετήσω ε, στο ελεκτικό συνέδριο ως αξιόπιστο μέλος και αφιέρωσα την ενέργειά μου ε, στο ε, έργο μου και στην εργασία μου ως ελεγκτής. Για τα επόμενα έτη θα παραμείνω σε αυτή την προσήλωση για να είμαι αξιόπιστο μέλος. Και θα ήθελα ε, να σας πω όταν εξετάσετε την υποψηφιότητά μου ότι μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα. Μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα και με τιμή θα απαντήσω στις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας, όχι μόνο σήμερα, ή δυνατόν και τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ζεντόφσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πένιγκ Μάια για την πολύ εντυπωσιακή εισαγωγή που κάνατε και θα ήθελα να σας ε, κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις αν μου επιτρέπετε. Πρώτα απ' όλα, αυτό που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στην ε, εισήγησή σας ε, σχετικά με το τι ακριβώς επιθυμείτε να κάνετε για τα επόμενα έξι χρόνια αυτό λοιπόν που είναι εντυπωσιακό είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Μήπως μπορείτε να μας ε, αναφέρετε τρία άλλα σημαντικά πράγματα, τι ακριβώς ε, προτίθεστε να προάγετε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, και πώς σκοπεύετε να γίνετε πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου ως ελεγκτής. Το δεύτερο θέμα αφορά στη συνεργασία. Βεβαίως όλοι λένε ότι πρέπει ε, να ε, συνεργαζόμαστε περισσότερο με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών, ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό που έχει εξίσου μεγάλη σημασία είναι πώς ακριβώς ε, προτίθεστε να συνεργαστείτε με τις εθνικές αρχές. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια. Ε, αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση και η τρίτη που θέλω να κάνω αφορά σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που είπατε. Αναφερθήκατε σε σύγχρονες τεχνικές ελέγχου. Τι ακριβώς εννοείτε με σύγχρονες τεχνικές. Μπορείτε λιγάκι να μας το εξηγήσετε, να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ε, δύσκολες ερωτήσεις. Θα μπορούσα να μιλάω για αυτά όλο το πρωί, αλλά θα είμαι πολύ σύντομο, γιατί ενδεχομένω να προσφερθεί και αργότερα η ευκαιρία να απαντήσω με περισσότερε λεπτομέρειε. Η πρώτη ερώτηση αφορά στην αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού συνεδρίου. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι πρέπει να μετακινηθούμε από ελέγχους οικονομικούς και ελέγχους συμμόρφωσης σε ελέγχους απόδοσης. Γιατί διαπιστώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα κονδύλια δαπανώνται όπως ακριβώς προβλέπεται, Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά το αποτέλεσμα ε, δεν έχει νόημα. Ε, Παραδείγματος χάρη λιμάνια χωρίς πλοία ή ε, αεροδρόμια χωρίς επιβάτες. Γι' αυτό λοιπόν η απόδοση είναι καθοριστική σημασία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο νομίζω ότι πρέπει να αναδιοργανώσουμε τους ελέγχους μας ε, και τη δήλωση αξιοπιστίας. Το δεύτερο θέμα έχει άμεση σχέση και μιλάμε για ε, περικοπή δαπανών. Μιλάμε για πάνω 60 εκατομμύρια και σας είπα το ποσό αυτό είναι υπερβολικό. Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε να ε, επιτυγχάνουμε δήλωση αξιοπιστίας ε, πολύ πιο φτηνά. Νομίζω ότι αυτό είναι απλό. Το τρίτο θέμα της ε, αποτελεσματικότητας έχει σχέση επαφές ε, με τον έξω κόσμο και αυτό αφορά ε, τα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια κατά τη διάρκεια της πρώτης εντολής μου εντατικοποίησα τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επισκέφτηκα την ΚΟΖΑΚ, την συνδιάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων άλλους, ε, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικά την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, αλλά και την Επιτροπή. Δηλαδή, ο διάλογος ε, με την Επιτροπή από την αρχή μέχρι το τέλος ενός ελέγχου είναι καθοριστική σημασία. και ε, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, τους δικαιούχους. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς δικαιούχους στα κράτη-μέλη για να ακούσω ε, ποιο είναι το πρόβλημά τους, πού ακριβώς υφίσταται. Η δεύτερη ερώτησή σας αφορά στη συνεργασία. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο με εθνικούς ανώτατους ελεγκτικούς φορείς, γιατί έχω διαπιστώσει ότι μερικές φορές ε, τα ε, πρότυπα των ε, ελέγχων καθιστούν δύσκολη τη συνεργασία και πολλές φορές τίτε το ερώτημα γιατί ακριβώς ε, να πρέπει να μας εμποδίζουν αυτά τα πρότυπα από μια επικοδομητική συνεργασία. Παραδείγματο χάρη προσπάθησα να συνεργαστώ ε, με τον φορέα μας ε, στην Ολλανδία, τον ομόλογό μας και τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών προσπάθησα να προκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προκαλέσω μια συζήτηση για ελέγχους με θέμα καινοτομία στον έλεγχο. Η καινοτομία είναι καθοριστική σημασία για τις εξελίξεις. Ε, όταν μιλάμε για καινοτομία στους ελέγχους, κατ' ουσίαν περί πρόκειται. Παραδείγματο χάρη, ε, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι τι είναι ακριβώς η απόδοση. Η κυρία Γεωργίευα αλλά και άλλοι επίτροποι έχουν ακριβώς εμπλακεί σε αυτό το θέμα του τι είναι η απόδοση. Αλλά για το ελεγκτικό συνέδριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ε, να μετρά την απόδοση με ρεαλιστικό τρόπο. Όχι, παραδείγματος χάρη, να συμμορφώνεται κανείς ε, με τους βασικούς δείκτες της απόδοσης, γιατί αυτό είναι απλό. Το δύσκολο είναι να αποδείξει κανείς στους Ευρωπαίους πολίτες ότι αυτό που κάνει η Ευρώπη έχει νόημα για την καθημερινή τους ζωή, για την καθημερινότητά τους. Ελπίζω να απάντησα ικανοποιητικά στις ερωτήσεις. Ο κ. Κουνάη, σκιώδης ηγητής ε, των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μπρένινγκ Μάια, και να σας ε, καλωσορίσω να σας ευχαριστήσω για τα τελευταία έξι χρόνια. Κατά την ακρόασή σας, πριν από έξι χρόνια, δεν ήμουν παρόν, δεν μπορούσα τότε και όμως ε, μελέτησα όλα αυτά που είπατε τότε και διαπίστωσα ότι είχατε αναφέρει δύο προτεραιότητες. Η μία προτεραιότητα ήταν ότι επιθυμούσατε να έχετε πιο στενή επαφή με τους Ευρωπαίους πολίτες και ως εκ τούτου θέλατε να ε, καταστήσετε λιγότερους περίπλοκους τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, θέλω να σας ρωτήσω, τα τελευταία έξι χρόνια ήταν επιτυχημένα και ε, ποιοι ήταν οι και ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε αν επανεκλεγείτε για τα επόμενα έξι χρόνια. Και έχω κι άλλο ένα ερώτημα. Ως ε, Ούγγρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ούγγρος Ευρωβουλευτής. Για μένα το κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χρηστή διαχείριση ε, των πόρων. Και όταν ένα κράτος μέλος ε, παραβιάζει αυτόν τον κανόνα και έχουμε δει τέτοια παραδείγματα, όταν δηλαδή μια κυβέρνηση δεν καταπολεμά τη διαφθορά και όταν η Όλαφ εγκαλεί ένα κράτος μέλος, κατ' ουσίαν υπήρξαν περιπτώσεις που τελικά ε, δεν έγινε τίποτα. Υπήρξαν ε, τέτοιες περιπτώσεις όπου μια κυβέρνηση παρέκαμψε τους κανόνες ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, τι μπορεί κανείς να κάνει για να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να ληφθούν νομοθετικά μέτρα ή μήπως ε, είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι φυστάμενοι κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε για αυτές τις ερωτήσεις ε, και εγώ σας ευχαριστώ. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Ε, πρόκειται για τον μέσο άνθρωπο, πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί του και πώς μπορεί να συνδέσει τα περίπλοκα του ελεγκτικού συνεδρίου με την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Τα τελευταία έξι χρόνια Ήμουνα σε επαφή με πάρα πολλούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν εμπλακεί σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ρώτησα ε, ποια είναι η εμπειρία σας με τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν υπάρχουν σφάλματα, πού οφείλονται αυτά. Και μάλιστα εστιάθηκα, εστίασα σε θέματα που ήταν σε μου, έρευνα και καινοτομία. Είχα πάρα πολλές επαφές στον τομέα της έρευνας και έτσι λοιπόν μπόρεσα να κατανοήσω τι είναι σημαντικό στην πραγματική ζωή. Και άλλο ένα παράδειγμα. Ε, τώρα είμαι εισηγητής για την απόδοση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξωτερικών οργανισμών και προσπαθώ να διατυπώσω την άποψη των ε, πολιτών. Στην κολονία η ε, ΕΣΑ είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με θέματα τεχνικά, με την ασφάλεια. Αυτό όμω αφορά τον Ευρωπαίο πολίτη. Ή η αίμα στο Άμστερνταμ για τα ιατρικά ε, είναι σημαντική για πάλι την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Προσπάθησα λοιπόν να έρθω σε επαφή με τον Ευρωπαίο πολίτη και να τον βάλω στην προμετωπίδα των ε, ερευνών μα. Το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, η ε, χρηστή διαχείριση, είναι πολύ σημαντική, γιατί ένα, μια βασική προπόθεση για την ευρωπαϊκή συνεργασία είναι η χρηστή διαχείριση. Όλα θα πρέπει να εντάσσονται μέσα σε αυτή την ευνομία. Παραδείγματο χάρη σε περιπτώσεις ε, διαφθοράς, η ευνομία, εφόσον αυτή παραβιάζεται, αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική απειλή για την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία. Άρα δηλαδή αυτό το θέμα είναι καθοριστική σημασία. Πιστεύω βέβαια ότι η αποτελεσματικότητα του να διαφυλάσσουμε το κράτος δικαίου, αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους θεσμούς. Παραδείγματο χάρη ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι αστυνομία. Εμείς δεν διεξάγουμε ανακριτικά αναλύσεις όμως εντοπίζουμε περιπτώσεις οι οποίες είναι προβληματικές, είναι ευαίσθητες και κατόπιν ε, παραπέμπουμε περαιτέρω το όλο θέμα, αλλά ε, τα κράτη-μέλη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Όλαφ, ο νέος Ευρωπαίος εισαγγελέα και η ΕΚΑ ε, θα πρέπει να προσπαθούν να συνεργάζονται στενά ε, για να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις οι οποίες αποτελούν απειλή για την χρηστή διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ο κ. Βογέ, ζητώ συγγνώμη. Ε, ε, λάθος πληροφόρηση είχα. Δεν πειράζει, κυρία Πρόεδρε. Α πάρει το λόγο η Μαρτίνα πρώτη. Euh, euh, ε, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, δουλειά που κάνετε εδώ και έξι χρόνια και η οποία αναγνωρίζεται για την ποιότητα από όλους εδώ στην αίθουσα και πρέπει να σας πω πως ε, διάβασα με πολύ προσοχή και τις ε, γραπτές σας ε, παρατηρήσεις, όπως επίσης και τα εισαγωγικά σας σχόλια και το γεγονός πως μιλάτε τόσο ξεκάθαρα για θέματα τα οποία μας αφορούν για να γίνουν πιο κατανοητά, πιο ευανάγνωστα, έτσι ώστε η δουλειά σας και η δικιά μας δουλειά υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι περισσότεροι από αυτούς φορολογούμενοι και είναι επίσης και αυτοί που μας εκλέγουν. Ως Ευρωβουλευτής είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος για το θέμα του πόσο κατανοητή πρέπει να είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοκατανόηση μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτών. Αυτό είναι απαραίτητο και γνωρίζουμε όλοι πως το πιο δύσκολο στην ζωή το να κάνει κανείς τα πράγματα πιο απλά. Σημείωσα το εξή. Εμείς, η καινούρια θητεία, για το θέμα, για το θέμα του πόσο ξεκάθαρα εκφραζόμαστε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Και πιστεύω ότι θα ήθελα ε, να, ε, και πιστεύω ότι μπορείτε και εσείς να μας περιγράψετε ε, ποιες δράσεις θα αναλάβετε τα επόμενα έξι χρόνια για να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που κάνατε αυτή την ερώτηση για το πόσο ξεκάθαρα ε, θα ονομάζουμε τα πράγματα. Κάποιοι ίσως το θεωρούν ε, όχι τόσο σημαντικό. Για μένα είναι κομβικό ε, ζήτημα για την δημοκρατία το να είναι όλα ξεκάθαρα σε επίπεδο αναφορών, συστάσεων, περιγραφών. Είναι λοιπόν στην καρδιά της προσπάθειας που κάνω αυτό το οποίο εσείς εντοπίσατε. Και βέβαια υπάρχει και ο κίνδυνος τον οποίο ε, αναφερθήκατε. Είναι περίπλοκη η Ευρώπη, είναι περίπλοκη η συνεργασία στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα της πολύ συχνά είναι περίπλοκα. Οπότε το να μιλάμε απλώς με απλά λόγια δεν είναι η λύση. Θα επανέλθω στην, ε, στον έλεγχο για το Horizon 2020 ο πραγματικός κίνδυνος ήταν ε, το πόσο περίπλοκοι ήταν οι κανόνες ε, τη στιγμή που προσπαθούσε κάποιος να εφαρμόσει το πρόγραμμα και αυτό δημιουργούσε και σφάλματα. Όταν ξεκίνησα αυτό τον έλεγχο, έστειλα μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντας «Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου την σχετική νομοθεσία». Και η απάντηση ήταν «Πώς δεν γίνεται, ελάτε να τα πούμε, γιατί θα σας πάρει ένα χρόνο ολόκληρο να κατανοήσετε αυτό το οποίο βρίσκεται στην νομοθεσία. Οπότε δεν θα πρέπει εμείς ε, να ασχοληθούμε μόνο με την περίπλοκη νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι το σχετικά συνηθισμένο. αυτό που πρέπει, και αυτό έγινε εκεί, είναι πως εντοπίσαμε πως κάποιες από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γεφυρώσει κάποιους περίπλικους κανονισμούς με καθημερινές πρακτικές και για να μπορέσουν να ε, χρησιμοποιηθούν αυτά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα κέντρα, η ψηφιακή πύλη, ε, όλα τα σχετικά, ε, η ενιαίοι e έλεγχοι, οι σημειωμένες ε, συμφωνίες ε, επιχορήγησης, όλα αυτά έγιναν για να διευκολύνουν τους χρήστες του Horizon 2020, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό, αλλά να συμβεί το ίδιο και στην εφαρμογή και στη λογοδοσία της χρήσης της ανάλυσης που έγινε των πόρων. Εγώ λοιπόν για το λόγο αυτό έχω προσθέσει μία λέξη η οποία για μένα είναι ε, σημαντική. Είναι η λέξη interface και γι' αυτό ε, έχω ε, προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους ε, διαδράσεις με ε, την νομοθεσία, με ε, τους πολίτες, γιατί πιστεύω πως υπάρχει, πάρα υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να δημιουργήσουμε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ της περίπλοκης νομοθεσίας και του κόσμου που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει αυτή την νομοθεσία, έτσι ώστε αυτή η συνεργασία να είναι ομαλή και χωρίς εμπόδια. Από τις άλλες πολιτικές ομάδες δεν βλέπω κανένα. Από τους προσένους. Α, η Μαρτίνα θέλει να κάνει ερώτηση. Α, ορίστε. Στη δεύτερη απόπειρα. Ε, ευχαριστώ. Ήμουν ε, τα περασμένα χρόνια σκιώδης εισηγήτρια και είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον Άλεξ Μπρένιγκ Μάιερ. Ε, είχαμε πολύ συχνά την ευκαιρία να συναντιόμαστε. Άλεξ, νομίζω ότι ο επαγγελματισμό σου ε, και γενικά ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεις τα πράγματα και τα γνωρίζεις είναι μοναδικός. Μπορείς εύκολα να συνδέεις τις λεπτομέρειες, όπως είδαμε στο Horizon, με τη συνολική εποπτεία. Και έχουμε κάτι κοινό οι δυο μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι η διαδικασία απαλλαγή είναι μια διαβίου μάθηση για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και το είδαμε στην περασμένη θητεία. Άρα, δεν θα σε εκπλήξει η ερώτησή μου. Ανέκαθεν ήθελες να ανανεώσεις, να καινοτομείς στην ε, διαδικασία του λογιστικού ελέγχου. Και στην απάντησή σου μας είπες ότι θα εξακολουθείς να στοχεύεις την απλούστευση ε, του λογιστικού ελέγχου. Πώς μπορεί λοιπόν να ανανεωθεί αυτός ο λογιστικός ε, έλεγχος και ε, να μην ανανεωθεί μόνο ο τρόπος με τον οποίο αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο ε, τα όσα έχει βρει στους ελέγχους, αλλά και η όλη διαδικασία. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που θα έχουμε να συνεργαστούμε και προβλέπω, προ, βλέπω συγγνώμη, σε αυτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εξίσου σημαντικό με το ορίζον 2020. Γι' αυτό το τελευταίο για την καινοτομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξέρω τι λέει η έκθεση και ε, ε, σας υπόσχομαι ότι θα σας βοηθήσει, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι δημόσια δεν μπορώ να σας αποκαλύψω το περιεχόμενό της. Ε, αυτό που ρωτήσατε για την καινοτομία στον έλεγχο και τη διαβίου μάθηση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή στη λογιστική στην Ευρώπη και στη λογοδοσία μάλλον στην Ευρώπη. Διότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει σε συνεργασία να αναζητήσουν έναν τρόπο να οργανωθεί η οικονομική ε, διοίκηση και ο έλεγχος ε, συμμόρφωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος του ελεκτικού συνεδριού είναι περιορισμένος μόνο. Ε, έχουμε την εποπτεία της ποιότητας ε, των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δεν μπορούμε σε επίπεδο δικαιούχων στα κράτη-μέλη να κάνουμε τόσο συστηματικούς ελέγχους και τόσο ε, πολλούς. Και αυτό είναι πρόβλημα και για τους ίδιους τους δικαιούχους το σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί με την ψηφιοποίηση του. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει τέτοιο στόχο να ψηφιοποιήσει την οικονομική της διοίκηση, ε, είναι καθημερινή δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λογοδοτεί ε, για όλες τις ε, δαπάνες και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Και σε μια δεύτερη φάση μπορεί να έρθει το ελεγκτικό συνέδριο να ελέγξει, να υποπτεύσει και να συμβουλεύσει το Κοινοβούλιο για οποιασδήποτε βελτιώσεις. Έτσι έχει λογική. Έχω πολλά πράγματα να σας πω, αλλά τώρα δεν μπορώ να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα είχα και εγώ μια καταληκτική ερώτηση σε σχέση με τις επιδόσεις, αυτό το performance. Δεν είναι εύκολο καθόλου να εκτιμηθεί αυτό. Να σας δώσω διάφορα παραδείγματα. Στο Βερολίνο έγινε ε, κάνανε μια διαδρομή ε, για τους μαθητές, για να μαθαίνουν την πόλη, Μα είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα διαρθρωτικά ταμεία να πληρώνει ε, ε, κυκλοφοριακά πάρκα, ας πούμε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής ε, για τους μαθητές μας. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Δεύτερη ερώτηση. Αρκετά συχνά χτίζονται διάφορα μικρά μουσεία για λόγους τουριστικούς σε φτωχές περιφέρειες ή σε περιφέρειες που υπάρχουν διαρθρωτικές δυσκολίες, το μουσείο τους μάρανε, ε, το, το, λαό εκεί της περιοχής, αυτό ένα μουσείο θα τους βοηθήσει. Είναι μικρά παραδείγματα, αλλά πραγματικά ε, δεν ξέρω κατά πόσο ε, είναι επίδοση αυτό το πράγμα και τελεσφορεί μια τέτοια δαπάνη. Εσείς έχετε δείκτες, δείκτες βασικούς και μας λέτε ότι δεν είναι αυτοί που προσφέρονται. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε αυτούς τους βασικούς δείκτες, τους key indicators, γιατί αν δεν έχουν καμία αξιοπιστία ως προς τις επιδόσεις, τι να τους κάνουμε. Είναι και λάθος επιλεγμένοι, λάθος σχεδιασμένοι και θα με ενδιαφέρει η απάντησή σας αυτό. Στα γερμανικά. Ε, τότε να πάμε και εμείς για εκμάθηση, όπως οι μαθητές στο Βερολίνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πιστεύω πως τα παραδείγματα που δώσατε ουσιαστικά φωτίζουν ένα από τα βασικά προβλήματα με τον ευρωπαϊκό προοικολογισμό και είναι το εξή. Και ίσως είναι και πολιτικά ευαίσθητο το θέμα, αλλά να σας πω ότι από τη σκοπιά του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου δεν υπάρχει καθόλου πολιτική πρόθεση, εμείς παρατηρούμε πως ένα πρόγραμμα δαπανών όταν βασίζεται στο να στέλνει χρήματα στα κράτη-μέλη ζητώντας από αυτά να καταθέσουν έργα, project, ε, τότε είναι σαν τα λεφτά να ψάχνουν project. Το αντίστροφο ε, ε, είναι η περίπτωση του Horizon 2020, όπου έχουμε τα project που ψάχνουν τα λεφτά. Πιστεύουμε λοιπόν, πιστεύουμε λοιπόν πως η πρώτη, το πρώτο σενάριο ε, ε, χρήματα ψάχνουν για project δεν είναι το πιο κατάλληλο. Και για το πάρκο αυτό το οποίο αναφερθήκατε και για το κομμάτι που αφορά τους μαθητές, το πρόβλημα είναι όντως το θέμα της απόδοσης των χρημάτων. Και εδώ ε, και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς στο Ελληνικό Συνέδριο θα πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα προόδου. Δηλαδή θα πρέπει η απόδοση να περιγράφεται μετά από διάλογο. Γιατί μπορεί κανείς να εντοπίσει ποια είναι η πρόθεση του προγράμματος και των κονδυλίων που θα δαπανηθούν. Δηλαδή ε, πώς πιστεύετε πως οι προθέσεις αυτές μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά. Και Όντω εξυπηρετούνται κάποιοι δημοκρατικοί στόχοι με αυτή τη διαδρομή την οποία ακολουθώντα οι μαθητέ θα διδαχθούν για τη δημοκρατία. Ναι, ενδεχομένω. Και ίσως αυτό να μπορεί να μετρηθεί ε, με δείκτες απόδοσης. Το Βερολίνο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτήσει αυτή τη διαδρομή η γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι λοιπόν μια ερώτηση αρκετά περίπλοκη. Πιστεύω όμω πω είναι σημαντικό. Γιατί θα να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πώ μπορούμε να την περιγράψουμε. Εκεί χρειαζόμαστε πρόοδο. Και πιστεύω πω και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Με κάθε project θα πρέπει να μπορούμε εμείς, η Ευρώπη, να εξηγήσουμε στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υλοποιούμε αυτό το project. Και αν μπορούμε να παρουσιάσουμε ε, μια κατανοητή εξήγηση, τότε εντάξει. Πολύ συχνά όμως έχουμε μπει σε μια καθημερινή δυναμική το ότι πρέπει να δαπανηθούν οι πόροι και βέβαια αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος. Άλλες ερωτήσεις έχετε? Όχι, από ό,τι βλέπω. Είναι πάρα πολύ πεπειραμένος ο υποψήφιός μας. Και σας κάλυψα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περιμένουμε το νέο υποψήφιο από τη Γαλλία. Έχουμε προβλέψει 45 λεπτά, λίγο περισσότερο χρόνο. Maintenant, c'est Φρανσουά Roger Καζαλά. Euh, Καλωσορίζουμε τον κύριο Φρανσουά Ροζέ Καζαλά. Σας καλωσορίζω θερμά και σας δίνω αμέσως το λόγο. Η δική σας εισηγήτρια είναι η κυρία Ισαβέλ Γαρθία Μουνιός. Κάθετε ξεβονίμων σας. Ε, σας δίνω αμέσως το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ ε, υποψήφιος της Γαλλίας για το ελεγκτικό συνέδριο. Ελπίζω πως θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, έτσι ώστε να ε, παρουσιάσετε την ε, γνώμη σας για την ε, υποψηφιότητά μου. Είμαι 62 χρονών, λέγομαι Καζαλά και από το 1979 είμαι μέλος της δημόσιας διοίκησης στη Γαλλία και από το 1981 και μετά δουλεύω στο Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Η καριέρα μου έχει μοιραστεί στα δύο. Σε δύο ίσα κομμάτια μέχρι σήμερα ήμουν ε, επιθεωρητής του Δημοσίου, μια και ήμουνα στο ελεκτικό συνέδριο της Γαλλίας και παράλληλα σε πιο επιχειρησιακό επίπεδο έχω και μια διεθνή διάσταση ευρωπαϊκή στη δουλειά μου. Είναι χρήσιμο για έναν ε, ελεγκτή να έχει επιχειρησιακή εμπειρία για να μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες και να κάνει ε, πραγματικούς ελέγχους. Σας παραπέμπω στο βιογραφικό μου για τις λεπτομέρειες του τι έχω κάνει στο ελεγκτικό συνάδελφο. Αν θέλετε μπορώ εδώ να επιμείνω σε μια διάσταση που είναι αυτή διεθνής και ευρωπαϊκή στα πλαίσια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Έξι χρόνια ήμουν στο Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, τρία χρόνια στην πρεσβεία στη Γερμανία και δέκα χρόνια στον Όσα, όπου το καθήκον μου ήταν να βοηθώ τις χώρες ε, υποψήφιας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας να στήσουν και να μεταρρυθμίσουν ε, τις δημόσιες δικήσεις τους πιο συγκεκριμένα για τα δημόσια οικονομικά που είναι ο χώρος μου. Ε, έκανα κάτι αντίστοιχο και για τους ελέγχους. Ε, για, τις, για τα αντίστοιχα ελεγκτικά συνέδρια των χωρών αυτών, αλλά και για τα Υπουργεία Οικονομικών που χρειάστηκε να στήσουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, δημοσιακού ελέγχου για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, ε, για τα προενταξιακά ταμεία και για τα ε, τα ταμεία αργότερα. Έχω λοιπόν διδαχτεί πολλά από αυτή την επαγγελματική ε, καριέρα και σε προσωπικό επίπεδο και ακολουθώ κάποιες αρχές οι οποίες κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ακολουθούνται από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο είμαι υποψήφιος. Η πρώτη αρχή, και δεν νομίζω ότι σα μαθαίνω κάτι καινούριο, είναι η ανεξαρτησία. Το πιο βασικό, η ανεξαρτησία ε, του θεσμού και των μελών που το υπηρετούν γιατί δεν μπορούμε να λαμβάνουμε οδηγίε από οποιονδήποτε, είτε για τον προγραμματισμό των εργασιών μα, είτε για τη χρήση και την επιλογή τη μεθοδολογία. Ε, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται η έκθεση. Δεν αποτε είναι δικαίωμα η ανεξαρτησία. Όχι, είναι υποχρέωση. Και δεν είναι αυτός σκοπός. Ε, δεν είναι προσωπική η αποστολή τους. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει για να προστατεύεται η καριέρα μας, αλλά η ανεξαρτησία αυτή θα πρέπει ε, να μην μας ε, κάνει ελεύθερους σκοπευτές. Ηλεκτρόνια που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, επιτρέψτε μου να πω. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συστήματος όπου ο ρόλος μας είναι σε ξεκάθαρη σύνδεση με τους υπόλοιπους ρόλους στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών και με το Κοινοβούλιο και θα πρέπει ο δημοκρατικός έλεγχος να γίνεται με τρόπο ε, σωστό, με σωστή συνεργασία και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με άλλα ε, ε, επίπεδα ελέγχου, για παράδειγμα, με τα μίδια Δηλαδή, θα προχωρήσω στο δεύτερο που είναι ο επαγγελματισμός. Δεν μπορούμε εμείς να εξηγούμε πως είμαστε ε, ανεξάρτητοι. Αν συνάμα αυτή την ανεξαρτησία δεν έχουμε και τον απαραίτητο επαγγελματισμό μέσω αυστηρών κανόνων που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και τη χρησιμότητα των ελέγχων μας. Ο επαγγελματισμός είναι η προστιθέμενη αξία του δικού μας ελέγχου, που είναι από τη φύση της μια κρίσιμη εργασία, όχι μόνο για να καταγγέλουμε τα σφάλματα και τα προβλήματα, αλλά για να βελτιώσουμε τη διαχείριση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εδώ και χρόνια εφαρμόζει αυτές τις αρχές και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της προώθησης που έδωσε και η δική σας επιτροπή ανάμεσα σε άλλους. Ακόμα όμως μένει πολύ πρόοδος να γίνει. Είναι οι σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα γιατί χωρίς ε, να διακυβεύεται η ανεξαρτησία και χωρίς να αλλάζει, θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να είναι σε συνεχή διάλογο με αυτά που ενδιαφέρουν τους ευρωβουλευτές και να προγραμματίζει αντίστοιχα την εργασία του. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στη σχέση με τα μίντια, ναι, αλλά η φήμη του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να ε, προστατευθεί ακόμα περισσότερο, να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί από τον Ευρωπαίο πολίτη έτσι ώστε να έχουμε και μεγαλύτερο κύρος. Επίσης, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ε, μεγαλύτερη ταχύτητα στις εργασίες μας και να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες της κοινή γνώμης έτσι ώστε να φωτίζουμε ακριβώς αυτά τα επίμαχα ζητήματα. Περισσότερη λοιπόν ευκρίνεια ε, να φωτίσουμε το τι συμβαίνει στις εργασίες μας έτσι ώστε οι συστάσεις μας να θέτονται σε εφαρμογή με έναν τρόπο που γίνεται κατανοητός και από τους πολίτες και από τους θεσμούς που ελέγχουμε. Δεν θα επιμείνω περισσότερο ε, για να μην μακρηγορήσω. γιατί θα πρέπει να δω πώς θα καταφέρω ε, να ε, μην σας κουράσω και παράλληλα να μην φανώ πως δεν γνωρίζω τα θέματα μου. Ε, ξέρω πως δεν είμαι ακόμα πολύ, απόλυτος γνώστης των όσων κάνω στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα κάνω κάθε προσπάθεια όμως για να σας ενημερώσω στα πλαίσια των όσων γνωρίζω και θα ακούσω τις ερωτήσεις σας για τις οποίες ήδη προημίου σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η συγκήτρια, κυρία Γκαρθία νιώθω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Καζαλά. Είμαι εγώ η ε, για την έκθεση του ορισμού σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πόσο σπουδαίο έργο η κυρία Ντανιέλα Μάρκ, η προκάτοχό σας, που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Και κρίμα ε, που αποχωρώντας η κυρία αυτή αλλάζει η ισορροπία του φύλου στο ελεγκτικό συνέδριο. Το Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε από τα αρμόδια όργανα και από το Συμβούλιο να ε, σέβεται την ισορροπία του φύλου στο ελεγκτικό συνέδριο. Δυστυχώς δεν καλύπτεται ε, η ποσόστοση των γυναικών. Το ξέρω ότι δεν φταίτε εσείς. Τώρα έρχομαι στα δικά σας θέματα. Διάβασα και μελέτησα το βιογραφικό σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι προφανές ότι έχετε και την εκπαίδευση και την εμπειρία ε, για τη θέση για την οποία σας προτείνουν. Διαβάζοντας όμως τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο μου γεννήθηκαν κάποιες επιφυλάξεις. Ήσασταν τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης ε, διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου της Υπουργού Περιβάλλοντος για λίγο χρόνο ε, και τα δύο αυτά πόστα είναι θέσει εμπιστοσύνη. Αλλά απαντώντα στην ερώτηση 5 λέγεται ότι δεν ήταν πολιτική καμία προηγούμενη θητεία σας, σε κανένα διορισμό σας και ήταν τελείως διοικητικής και τεχνικής φύσεως. Μα δεν θεωρείτε ότι οι θέσεις αυτές είναι πολιτικές ως προς τον διορισμό τους. Ε, περάσατε από πολιτικό γραφείο, ιδιαίτερο γραφείο Υπουργού βέβαια για σύντομο διάστημα. Γιατί γυρίσατε γρήγορα μετά στο ελεκτικό συνέδριο. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχουν μέλη του ελεκτικού συνεδρίου που διατέλεσαν εδώ ευρωβουλευτές και ήταν μέλη πολιτικών κομμάτων, ιδιαίτερα κάποιους που έχω υπόψη μου. Και υπάρχει απέτηση ε, για το ελεκτικό συνέδριο πάντες να είναι ανεξάρτητη. Και το πιστεύουμε ότι είναι. Εσείς αναφερθήκατε στην ανεξαρτησία και όχι μόνο σε αυτό. Στην απάντησή σας στην ερώτηση 7 λέτε ότι είναι σκόπιμο να απέχει κανείς από δράσεις, να λαμβάνει δημόσια θέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποψία ε, έλλειψη ανεξαρτησίας. Τι σημαίνει αυτό. Δεν θα πρέπει μόνο να είσαι ανεξάρτητος, αλλά να φαίνεσαι κιόλας. Αυτό μου φαίνεται πολύ καλό, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σωστό, αλλά στην πράξη τώρα αν θέλετε να το εφαρμόσετε, αλλάξτε ε, το προφίλ σας στο facebook και κάντε το ιδιωτικό και όχι δημόσιο γιατί τώρα μπορούν οι πάντες να διαβάζουν τις απόψεις σας. Ε, έχετε οριστεί υποψηφίους για μια πάρα πολύ σημαντική θέση στην Ευρώπη και ορισμένες δημόσιες δηλώσεις σας μπορεί να γεννήσουν υποψίες έλλειψη ανεξαρτησίας και τα αφήνω εδώ. Ε, σε ό,τι αφορά για την ανεξαρτησία μας βεβαιώνεται απαντώντας στην ερώτηση 13 ότι είστε ανεξάρτητο σε σχέση με το κράτος μέλος σας θα μπορούσατε να μας πείτε το ίδιο και για την πολιτική απόχρωση των κυβερνήσεων. Ας πούμε τι γίνεται με τις εκθέσεις για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως του κόμματος που κυβερνάει. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία που εσείς θα φέρετε ε, στο ελεγκτικό συνέδριο. Ποια θα ήταν οι προτεραιότητές σας ως ε, μέλος. Τι πιστεύετε για τις διαφορές, τις τεχνικές και πολιτικές ε, των νυν ελεγκτών. Η συνεργασία ε, με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και τους ομολόγους έχει αυξηθεί από την ίδρυση του ελεγκτικού συνεδρίου από την σκοπιά ενός εθνικού ελεγκτικού συνέδριου θεωρείτε ότι είναι πια βέλτιστη η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή χωράει βελτίωση. Και προς την κατεύθυνση αυτή ποια μέτρα θα προτείνατε. Και όσο για τις ε, συνεργασίες, απαντώντας στην ερώτηση 15, ε, λέτε ότι καλή την πίστη θα πρέπει να συνεργάζεται το συνέδριο με το Κοινοβούλιο. Δεν θα μπορούσε ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση να ελέγχετε, να επιλέγετε κάποια θέματα που ελέγχεται που να είναι θέματα που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο. Ε, το ξέρω ότι θέλετε να συνεννοήσετε με το Κοινοβούλιο, ε, αλλά το ελεκτικό συνέδριο ε, υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του και είναι πολύ σε αυτή η δυνατότητα που έχει να επιλέγει τα θέματα, όπως και το γαλλικό άλλωστε. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει όλο και περισσότερη έμφαση ε, στην εκπόνηση ειδικών εκθέσεων χωρίς βεβαίως ε, να υποτιμά, να υποβαθμίζει το γενικότερο έλεγχο. Ποια είναι η άποψή σας ε, για ε, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Γνωρίζετε πώς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι από την προηγούμενη εμπειρία σας. Ε, κάνατε τέτοιους ελέγχους στο Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Και για να τελειώνω, παρόλο που έχω και άλλες ερωτήσεις, θα κάνω τελευταία, γιατί βλέπω την Πρόεδρο ήδη να μου κάνει νοήματα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερη τάση να ελέγχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια περισσότερο από κάποια άλλα. Στη Γαλλία τι γίνεται. Χρειάστηκε να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια θητείας σας για κάποια υποψία απάτης ή διαφθοράς. Κάνατε ελέγχους πολλούς ε, για τα διορθωτικά για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα σας. Σταματώ εδώ. Το ξέρω ότι έχω κάνει πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε όμως παρακαλώ τους συναδέλφους να δώσουν την ευκαιρία να απαντάει και ο υποψήφιος. Αν τον βομβαρδίζετε με τις ερωτήσεις είναι λίγο δύσκολο. Ήταν πολλές αλλά και πολύ καλές οι ερωτήσεις ε, και θα σας παρακαλούσα τώρα κύριε Καζαλά να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε. τα σημείωσα, αλλά αν δεν τα έχω σημειώσει όλα, διακόψτε με και υπενθυμίστε μου ε, τα λεγόμενά σας. Το πρώτο ήταν μια διαπίστωση, ναι. Δεν ευθύνομαι. Είμαι όντως άνδρας υποψήφιος. Τώρα για να επανέλθω στο ουσιαστικό θέμα που θέσατε για τη θέση μου σε γραφείο υπουργού. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ παλιό. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώ ήταν, πριν από 25 περίπου χρόνια. Νομίζω παραγραφή πια για τέτοιου είδου θέματο. Ε, Τώρα, επιμένω, δεν υπήρχε καμία πολιτική χρειά στην ε, θέση αυτή. Βεβαίω έπρεπε να έχω την εμπιστοσύνη του Υπουργού, αλλά δυστυχώ στη Γαλλία είναι έτσι το σύστημα όπου οι τεχνοκράτε, στου οποίου ανήκω, ε, ε, πάντοτε την χάνουν τη εμπιστοσύνη των Υπουργών. Ίσως αυτό είναι αρνητικό, ίσως να έχει κάποιο πολιτικό κόστος. Εμείς με ρωτήσατε γιατί έφυγα από το γραφείο του Υπουργού γιατί κάποια στιγμή προτίμησα να απομακρυνθώ ε, κοινή συμφωνία από τον Υπουργό ε, μετά από μια ε, κυβερνητική αλλαγή και γιατί είχα οικογενειακούς λόγους που με οδήγησαν να επιστρέψω στο ελεγκτικό συνέδριο. Για το προφίλ μου στο facebook, σας ευχαριστώ. Αυτό σκεφτόμουν ερχόμενος και σας υπόσχομαι Σας υπόσχομαι να είμαι πολύ προσεκτικός και βεβαίως ε, ε, σας εκτιμώ για την προσοχή με την οποία αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα. Για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ίσως δεν πρόλαβα να τα σημειώσω όλα. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος που κατάλαβα ε, τι ακριβώς σημαίνει ε, τεχνικό και πολιτικό προφίλ και αν είναι η πολυμορφία των τεχνικών προφίλ και αν αυτό είναι ευκταίο ε, όχι, για μένα ναι. Για παράδειγμα, στο Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουμε νομικούς, έχουμε οικονομολόγους, έχουμε λογιστές, έχουμε μηχανικούς. Άρα ναι, πολυμορφία, διεθνής εμπειρία Μόλις ήρθε ένα συνάδελφος που ήταν διπλωματικός στο παρελθόν και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το ότι έχουμε αυτά τα διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ, αν και θα πρέπει βεβαίως όλοι να γνωρίζουν τα βασικά του καθήκοντα, που είναι η εξέταση των λογαριασμών. Αυτό για μας θεωρείται πλεονέκτημα. Και είναι υπέρ μας ότι υπάρχει αυτή η πολυμορφία Πρώτον, γιατί υπάρχουν πολλαπλές απόψεις και δεύτερον, γιατί μπορούμε να σταθούμε σωστά ενώπιον αυτών που ελέγχουμε. Εγώ, για παράδειγμα, για 7 χρόνια είχα τις μεταφορές και όταν πήγαινα στο Υπουργείο Μεταφορών με συνάδελφο που ήταν μηχανικός, αισθανόμουν πιο άνετα. Δεν θα έλεγα πιο άνετα. Ε, αισθανόμουν πως ε, με σέβονται περισσότερο ε, και σεβόντουσαν περισσότερο το θεσμό τον οποίο εκπροσωπώ ακριβώς επειδή είχαμε και αυτή τη γνώση. Εσείς είπατε πως ε, για να κάνουμε αυτό το performance audit θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες αρμοδιότητες και όχι μόνο οι νομικές, οικονομικές ή λογιστικές. Ναι, το ελεγκτικό γαλλικό ε, συνέδριο εδώ και χρόνια έχει τέτοιου είδους δραστηριότητα και παρόλο που καμιά φορά και μπορούμε να βάλουμε σε αυτή την κατηγορία τον έλεγχο το οποίο είχα το συντονισμό ε, για τα τρένα υψηλής ταχύτητας ε, στη Γαλλία δεν ξέρω αν ήταν νομικά τα θέματα, δεν ξέρω αν ήταν θέμα λογαριασμού, ήταν εντάξει, αλλά ε, είδαμε το κατά πόσο αυτά τα τρένα υψηλής ταχύτητας ήταν η κατάλληλη περιβαντολογική και οικονομική απόκριση στο σημερινό πλαίσιο που είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο έγιναν αυτές οι επενδύσεις ε, πριν από 25 χρόνια. Αυτό ήταν λοιπόν, αυτό ήταν ένας από τους φακέλους μου, για παράδειγμα. Και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα επανέλθω. Τώρα, συνεργασία πιο συγκεκριμένα μεταξύ του Εθνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκού. Η ε, μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί. Θυμάμαι την εποχή όπου επέστρεψα στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από τη θητεία μου στο Υπουργικό Γραφείο, συμμετείχα σε ομάδες εργασίας που ήταν υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή πάλι πριν από 25 χρόνια, και τότε ε, ήταν έτσι κάπως παράξενο. Πολύ λίγοι ενδιαφερόντουσαν, και δεν ήταν και πολύ δραστήριο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα ευτυχώ τα πράγματα έχουν αλλάξει και μπορώ να πω και είναι πραγματικότητα και τουλάχιστον για το Γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο ε, και εσείς ε, μιλήσατε για τη συνάδελφο που ήταν ε, υπεύθυνη για τα θέματα αυτά στο ε, Γαλλικό Ελληνικό Συνέδριο και μετά πήγε στο Ευρωπαϊκό, να σας πω πως είναι λοιπόν υπεύθυνη για την ε, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ μας. Ε, δουλέψαμε πολύ καλά μαζί και εκτός από αυτά που είπατε εσείς, θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα συνεργασίας. Πρώτα απ' όλα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας και για τις μεταφορές πιο συγκεκριμένα κάναμε τακτικές συναντήσεις το δικό μου τμήμα με το αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ανταλλάσσαμε ε, προγράμματα, βασικές διαπιστώσεις, ε, μεθοδολογίες και ο έλεγχος αυτός Μας κάλεσαν δημόσια στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να παρουσιάσουμε τον έλεγχο μας αυτό και νομίζω ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κάναμε και αλλού και ήταν σημαντικό που έγινε και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πιο πρόσφατα, γιατί έχω δύο χρόνια που δεν είμαι στι ε, στο, μεταφορές αλλά στα δημόσια οικονομικά, εδώ είναι κάπως αντίστροφη η κατάσταση. Προηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο. Εμείς τώρα κλείνουμε έναν ε, έλεγχο για τα μεγάλα ε, επενδυτικά σχέδια στην Ευρώπη, αυτό το οποίο ονομάζεται πακέτο Juncker. Στη Γαλλία ήρθαμε αμέσως σε επαφή με τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ξέραμε ότι είχαν κάνει και έκθεση ε, για τα πρώτα μέτρα για το πακέτο Juncker και επίσης είχαν καταθέσει γνωμοδότηση για την ε, επέκταση αυτού του σχεδίου. Εμείς λοιπόν χρησιμοποιήσαμε την πραγματογνωμοσύνη τους και αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα για ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο και το οποίο είχε τέτοιου είδους δείκτες απόδοσης, ήταν ένα είδος ε, αξιολόγησης απόδοσης Προσωπικά δεν συμμετείχα στον έλεγχο ε, για το πώς ε, εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια στη Γαλλία. Ξέρω πως έχουν γίνει και για τα γεωργικά κονδύλια και για τα διαστροτικά ταμεία. Για το πώς υλοποιούνται δηλαδή, το έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Δεν θα αναφερθώ για το ε, ναι, στον έλεγχο για το σχέδιο Juncker. Είναι διαφορετικό το θέμα. Ήταν ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία τα οποία συνδυάζονται ε, με τα, με τα κλασικά ταμεία και πώς αυτά χρησιμοποιούνται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να σας πω πως όταν ήμουν στις μεταφορές είχαμε την σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ Λιών και Τωρίνου, ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και για τη Γαλλία και για την Ιταλία αλλά και για την Ευρώπη, μια και το 30% του διεθνούς τμήματος θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε και άλλα θέματα παρόμοιας φύσης. αν χρειάστηκε να έρθω σε επαφή με υπόνοιες απάτης, πρέπει να σας πω όχι στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά για εγχώριες, για εγχώριες υποθέσεις, για διεθνείς υποθέσεις, ναι, είχαμε και διαφθορά, είχαμε και απάτη. Νομίζω ότι δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά στις περισσότερες από αυτές νομίζω έχω δώσει μία απόκριση και αν υπάρχουν κενά υπενθυμίστε τα σας παρακαλώ πολύ. Α, για τις προτεραιότητες. Μίλησα λίγο για τις προτεραιότητες. Για τις κλαδικές, για παράδειγμα, προτεραιότητες. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω τώρα. δεν είχαμε πληροφορίες ακόμα για το ποια, ποιος κλάδος θα αναλάβω. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για προτεραιότητες. Δύο πράγματα μπορώ να πω για τα όσα γνώριζα, γιατί και εγώ όταν ήμουν στον ΩΣΑ λάμβανα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι το πρόγραμμα ΣΥΓΜΑ, το οποίο υπάρχει ακόμα και το οποίο χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμουνα λοιπόν σε... Ήμουν δικαιούχος εκεί σε κονδύλια και πρέπει να σας πω πως χρησιμοποιήθηκαν στις, ε, υπο... στις υποψήφιες χώρες και εκεί νομίζω ναι, κάποιες προτεραιότητες χαράχθηκαν αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα. Είναι ένας πολύ ιδιάζων χώρος. Αντίθετα πρέπει να σας πω πως έχω πιο γενικές προτεραιότητες. Το είπατε κι εσείς, συνεργασία μεταξύ των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων, μια και προέρχομαι από εθνικό ελεγκτικό συνέδριο. Και ίσως έχω και είμαι πιο κατάλληλος από άλλους για να σκεφτώ τα θέματα αυτά και να δω πού μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας και να τη θέσουμε σε εφαρμογή και δεύτερον σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω πως έχετε δίκιο. Δεν πρόκειται εμείς να παραδώσουμε την ανεξαρτησία μας. θα ήμουν ο πρώτος ο οποίος ε, θα προσπαθούσα να παραμείνω σε ίση απόσταση μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, χωρίς όμως να απομονωνόμαστε, γιατί καμιά φορά με πολύ συστηματικό και ίσως παθολογικό τρόπο υπερασπίζεται κανείς την ανεξαρτησία του. Θα πρέπει ίσως λοιπόν να σεβαστούμε την αυτονομία των μεν και των δε, να το πούμε έτσι, και να οργανωθούμε με έναν τρόπο που θα υπηρετεί το στόχο της συνεργασίας που θα είναι αποτελεσματική. Για πολύ χρόνο το, ο θεσμός στον οποίο ανήκω αντιμετώπιζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάποια ενδεχομένως έλλειψη εμπιστοσύνης. Υπάρχουν λόγοι. Ξέρετε ποια είναι η νομική φύση του Γαλλικού όπως και του Ισπανικού Ελεκτικού Συνεδρίου. Εκεί αντιμετωπίζαμε το Κοινοβούλιο κάθε φορά ως θεσμό που δεν είναι ε, παρόμοιος με το δικό μας και που μπορεί οριακά να θεωρηθεί πως είναι και σε αντίθετη πορεία από αυτή που βρισκόμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, θυμάμαι τον Φιλίπ Σαγκά που ήταν και πρόεδρος της Βουλής και ήταν και ο πρώτος πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και αυτή η διπλή αρμοδιότητα του επέτρεψε να δει τα πλεονεκτήματα που θα έφερνε η πιο στενή συνεργασία με την ε, Βουλή και τη Γερουσία στη Γαλλία. Και έγινε αυτό με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Αλλά ξεκινούσαμε από πολύ ε, χαμηλή βάση, μηδενικές επαφές και φτάσαμε σε κάτι το οποίο τελικά είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ αποτελεσματικό. Εντάξει, δεν έχω αυταπάτες για την ποσότητα της προσθέμενης αξίας που θα φέρει αυτό. Μικρή θα είναι, θα πρέπει βέβαια οι ευρωβουλευτές να ενδιαφέρονται για το έργο μας, θα πρέπει εμείς να είμαστε στη διάθεσή τους, αλλά νομίζω πως είναι απαραίτητο. Αυτά. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ich glaube, sehr umfassend Νομίζω ότι δεν φοβηθήκατε να απαντήσετε. Μπας περιπτώσει, αν θέλει κάποιος μπορεί να υποβάλει και άλλες συμπληρωματικέ ερωτήσεις. Επόμενος ο κύριος Ζεντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το μέλος του ε, ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να είναι λακωνικό ένα μέλος και να μην θέλει τώρα 15 ολόκληρα λεπτά για να απαντήσει σε μία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ πρώτη ερώτηση. Τι ακριβώ επιθυμείτε, τι θέλετε να αλλάξετε όσον αφορά τους ελέγχους. Ενώ την απόδοση των ελέγχων. Ε, τι σημαίνει ο για τον πολίτη. Δεύτερη ερώτηση αφορά τις ε, πολύ καλές σας γνώσεις για το πώς λειτουργούν οι έλεγχοι. Αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε πώς επιθυμείτε να συνδέσετε τους εθνικούς με τους ευρωπαϊκούς ελέγχους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα, ας πούμε, στους ε, γαλλικούς ελέγχους ε, και τους ευρωπαϊκούς ελέγχους. Και η τρίτη ερώτηση αφορά περισσότερο στις ε, επιθυμίες σας, δηλαδή είπατε ότι ε, δεν ξέρετε ακριβώς σε ποιο τμήμα ε, θα ενταχθείτε ή που θα πάτε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς τμήμα προτιμάτε. έχετε υπόψη κάποιο συγκεκριμένο τμήμα, τι ακριβώς κάνουν, ποιες είναι οι του. Ε, Μήπω έχετε υπόψη σας αν υπάρχει ένα τμήμα το οποίο να εστιάζεται περισσότερο ε, σε θέματα με τα οποία ασχοληθήκατε κατά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Βουλευτά, μία παρατήρηση ε, μακρηγόρησα για να απαντήσω, αλλά δεν απαντούσα σε μία ερώτηση, απαντούσα σε 15 ερωτήσεις. Εντάξει, τούτου λεχθέντος έχετε δίκιο, αλλά ακόμα δεν είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και ίσως έχω την τάση να μακρηγορώ λίγο και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. Ε, πώς να κάνουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου πιο προσβάσιμα και εύληπτα για τους πολίτες, αν κατάλαβα καλά την πρώτη σας ερώτηση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Είπα την πολιτική επικοινωνία πρώτα απ' όλα, η οποία έχει βελτιωθεί πολύ στο ελεκτικό συνέδριο νομίζω. Το είδα διαβάζοντας τι ειδικέ εκθέσεις στον σχετικό κατάλογο. Στο παρελθόν ήταν ε, ε, μια λιτανία έτσι αρκετά βαρετή. Ε, τώρα εστιάζουν στη συγκεκριμένη έκθεση. Βεβαίω παραμένουν εκθέσει αυτέ πάρα πολύ τεχνικέ και είναι γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, μπορεί λίγο. Πώ να το πω τώρα. Ορίστε, χάνω και τα λόγια μου. Ε, και εγώ, μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ το πιο ε, αγαπημένο τους ανάγνωσμα αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν απλούστευση, διευκρίνηση, ε, Περιορισμό σίγουρα το, της έκτασης των εκθέσεων, ε, αποφεύγοντας να χάσουμε την ουσία και την αυστηρότητά τους. Είναι δύσκολο αυτό και εμείς έχουμε πρόβλημα ε, για να κάνουμε τις εκθέσεις μας πιο ε, ευληπτές και ευανάγνωσες χωρίς να χάσουμε την επαγγελματική ποιότητα. Και όταν κάποιος κάνει λογιστικό έλεγχο και καλείται να κάνει έκθεση στη συνέχεια, πάντα ε, χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες αποχρώσεις, κάποιες παραμέτρους και αυτό κινδυνεύει να θολώνει το μήνυμα. Αλλά είναι περίπλοκες οι καταστάσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει αυτό. Ε, από τη μια υπάρχει η ε, επιθυμία να είμαστε πιο σαφείς και πιο ευανάγνωστοι, από την άλλη η υποχρέωση να διατηρούμε την ε, μεθοδολογία μας, την αντικειμενικότητά μας. Αυτό που έχει σημασία είναι να καλές συστάσεις για να είναι χρήσιμες και στα ε, όργανα που ελέγχουμε έτσι ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν πάντα προς το συμφέρον των πολιτών. Αυτή η διαδικασία είναι κάπως έμεση, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Να ενημερώνουμε τους πολίτες και να τους βοηθούμε να λαμβάνουν ε, θέση ε, στη δημόσια συζήτηση, αλλά κάνουμε και συστάσεις οι οποίες τελικά θα επιτρέψουν να βελτιώνεται η διαχείριση και η εκτέλεση των προϋπολογισμών στο κάτω-κάτω είναι και χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Ακόμα και αν είναι έμεσο αυτό το μέσο, βοηθάει να βελτιωθεί η κατάσταση. Σύνδεση τώρα ε, των εθνικών θεσμών με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Νομίζω ήδη έχουν γίνει πολλά. Μπορούμε να προχωρήσουμε και παραπέρα, αλλά αυτό εξαρτάται και από τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια, όχι μόνο από το ευρωπαϊκό όσο καλή ε, θέληση και να έχει. Εμείς τι κάνουμε. Και πάλι αυτό διαφέρει από ελεκτικό συνέδριο από χώρα σε χώρα. Μπορεί να χρειάζεται να γίνεται πιο συστηματικά. Έχουμε ε, συνεδριάσεις ανταλλαγής πληροφοριών. Είτε συνολικά μία ετήσια ας πούμε συνεδρίαση ε, για το σύνολο των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν και είναι στην επικαιρότητα και από την άλλη υπάρχουν και επιμέρους. Όπως σας ανέφερα, είχα τις μεταφορές εγώ για σειρά ετών. Είχαμε τουλάχιστον κάθε εξάμεινο συνεδρίαση ειδική για τις μεταφορές. Άρα έχουμε επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό είναι το ένα. Βέβαια συζητούμε επίσης και ε, τα προγράμματα εργασίων μας σπανιότερα ε, για να βεβαιωθούμε ε, να μην υπάρχουν επικαλύψεις πάρα πολλές που είναι σπάνιο όπως είπα και να δούμε τι λένε οι συνθήκες και ποιες δυνατότητες έχουν τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να ε, πλαισιώνουν, να συνοδεύουν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όταν έρχεται να κάνει επιτόπιους ελέγχους. Στην αρχή το κάναμε σπανιότατα, ε, ε, τώρα όλο και περισσότερο, χωρίς αυτό να είναι συστηματικό. Και αυτό αποδεικνύει ότι εμπιστευόμαστε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το τρίτο που είναι ίσως πιο δύσκολο να υλοποιηθεί και εξ όσων γνωρίζουν δεν έχει ακόμα πλήρως οριστικοποιηθεί είναι το να κάνουμε ελέγχους όχι ακριβώς κοινού, αλλά παράλληλους. Είναι κοινό το θέμα και η μεθοδολογία ε, συγκρίνεται ε, και αντιπαρατίθεται ας πούμε και συγκρίνουμε και τα αποτελέσματα. Ξέρω ότι αυτό έχει γίνει σε κάποιες χώρες, αλλά για να μην πω καμιά βλακεία, ε, δεν θα την κατανομάσω. Νομίζω η πρόεδρος μίλησε για μια χώρα ε, που έχουν μεγάλη, μάλλον οι κυρίες ηγήτρες, συγγνώμη, ε, για χώρες που κάνουν περισσότερους ελέγχους στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό γίνεται πιο εύκολα γιατί υπάρχει ένας φυσικός συντονισμός ελεγκτικού και εθνικού εκάστοτε ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ποιο τμήμα θα πάω. Ε, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή. Είναι λίγο λεπτή. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον πρόεδρο, τον κύριο Λένε, ε, το, το οποίο ακρόαση ακολουθεί ε, για τα θέματα αυτά. Έχω ένα μικρό πρόβλημα να απαντήσω. Το τμήμα που ασχολείται με τα ταμεία συνοχής και τα διορθωτικά ταμεία είναι πάρα πολύ δημοφιλές ε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πάρα πολύ ε, πολύπλευρο. Επίσης, τίνω να πιστεύω ότι η παρελθούσα εμπειρία μου θα μπορούσε να με οδηγήσει αρκετά φυσικά και ε, σε θέματα μεταφορών ή διεθνούς συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, κάτι που αποκλείεται κατά τη γνώμη μου, παρόλο που θα μου άρεσε να ασχοληθώ, είναι ό,τι έχει σχέση με την Τραπεζική Ένωση, τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με αυτό ασχολούμαι αυτή τη στιγμή. Ακόμα μαθαίνω, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω και αισθάνομαι ότι έχω κάποια επάρκεια για να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το Renew Europe, ο κύριος Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Καζαλά και για την παρουσίασή σας, αλλά και για τις γραπτές σας παρατηρήσεις που μας διαβιβάσατε εκ των προτέρων. Έχω ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή μας ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει όλο και περισσότερο να αναλύει την απόδοση της επιδόσης. Θα πρέπει να πιάνει τόπο το κάθε ευρώ και με τρόπο ευφυή να δαπανάτε και όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό, σε, με βάση αυτά που γνωρίζετε. Ε, Πώς αξιολογείται τη σημερινή δραστηριότητα του ελεγκτικού συνεδρίου και τι πιστεύετε για τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιεί μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στους διάφορους λογιστικούς ελέγχους. Στην απάντησή σας μιλάτε για χρηστή διαχείριση και ε, γερή ε, ε, δημόσια διακυβέρνηση τι εννοείτε, ποια είναι αυτή η δημόσια διακυβέρνηση και πού ε, βλέπετε να χωράει η βελτίωση ε, στα ευρωπαϊκά θέματα. Και τέλος, πάντα στο φάκελό σας επιμένετε πάρα πολύ στη διαφάνεια. Τι θα πρέπει να κάνουμε κατά την άποψή σας για να βελτιώσουμε αυτή τη διαφάνεια και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ακαιρεότητα των οργάνων και η λειτουργία τους. Ευχαριστώ. Ε, πώς να είμαι σύντομος τώρα. Δύσκολο θα είναι. Merci, Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Οι ερωτήσει σα είναι πάρα πολύ σχετικές και άπτονται θεμάτων που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και θα μιλήσω τώρα για την απόδοση. Θα χαρώ να σας απαντήσω γιατί αναφέρθηκα στην εποχή ε, που ήμουν σταζιέρ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγγνώμη, με συγχωρείτε, που χρησιμοποιήθηκε ως τεχνικός εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες ε, υποψήφιες για ένταξη. Και τότε είχαμε αναρωτηθεί το εξή: Ποια είναι η χρήση των δράσεων που χρηματοδοτούμε και ποιος είναι ο πιο χρηστός τρόπος για να εξασφαλίσουμε ε, τις κατάλληλες δράσεις και όχι άχρηστες, θα το πω έτσι, βλαβερές ή αδιάφορες. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είδαν να χρηματοδοτούνται δράσεις ε, οι οποίες δεν ήταν ε, κάτι το ιδιαίτερο. Μιλώ για συμβουλευτική, για παράδειγμα, που δεν κόστισε πολύ, αλλά ποσά τα οποία δεν ήταν αμελητεία και με ενοχλούσε το ότι είχαν, είχαν χρηματοδοτηθεί ακολουθώντας τους σωστούς κανόνες, αλλά για να πληρωθούν τσαρλατάνοι. Δεν βοηθούσε αυτά τα κράτη τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτήν την τεχνική βοήθεια. Οπότε, ε, ε, και θα ήθελα ε, να ε, με ακούσετε. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εξετάσαμε την κανονικότητα. Ε, που δεν είναι. Ήταν απλώς μία κρίση προσωπική για τη χρησιμότητα, όχι. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει ε, και τους πόρους που έχει, αν δεν κάνει ελέγχους οι οποίοι αποδίδουν στην πραγματικότητα. Για τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει αυτή τη δουλειά με τους δείκτες για την απόδοση, πρέπει να παραδεχθώ πως δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν κατέχω επαρκώς το θέμα. Εγώ γνωρίζω καλύτερα τα εμπορικά θέματα και νομίζω ότι ε, στο σημείο της απαλλαγής θα πρέπει να εξετάσω όλα τα θέματα αυτά με κριτικό πνεύμα, αλλά ε, θεωρώ πως θα υπάρχουν και δείκτες απόδοσης του ίδιου του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι συστάσεις, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί. Ας είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση των δικτών. Γιατί καμιά φορά συγχαίουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα με λιγότερο σαφή που δεν είναι απαραίτητο αντιπροσωπευτικά ε, για να κρίνει κανείς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα ενός θεσμού. Αλλά σας παρακαλώ πολύ ε, εδώ να με κρίνετε με επίοικια τώρα για την δημόσια διαχείριση και τον έλεγχο. Και αυτό πάλι μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές, γιατί όταν ήμουν στον ΩΣΑ και είδα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είδα πως θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη εστίαση σε συγκεκριμένο χώρο ε, της δημόσιας διοίκησης και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα, ε, τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ ενδιαφέρον για όσους χρηματοδοτούσαν και συγχωρέστε με τώρα που μπαίνω σε φιλοσοφικά χωράφια, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν τμήμα ενός συστήματος. Συστήματος που χαρακτηρίζεται από αυστηρή ιδιοντολογία, αυστηρή ακυριότητα, που θα προστατεύει από πολιτικές πιέσεις τους δημόσιους λειτουργούς, που θα έχει ποιοτική πρόσληψη, ποιοτική εκπαίδευση αυτών και αυτά τα στοιχεία είναι ανεξάρτητα από τα στοιχεία του ελέγχου, αλλά παρόλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα κατά τη δική μου γνώμη γιατί ένας έλεγχος δεν είναι μόνο τεχνικά καλός είναι επίσης καλός γιατί έγινε με τον κατάλληλο επαγγελματία που παρουσιάζει τα απαραίτητα εχέγγυα μέσω καριέρας και που γνωρίζει τα θέματα δημόσιας διοίκησης καλύπτει πίστη δε επειδή όλα αυτά είναι στο πεδίο της εντολής τους. Letzte Frage Dobré eh, eh, Σας eh, καλημερίζω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω έναν υποψήφιο ο οποίος ε, έχει εμπειρία από το δημόσιο χώρο και είναι και πολιτικά ανεξάρτητος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα. Έχω λοιπόν ένα πιο γενικής φύσεως ερώτημα, το οποίο δεν αφορά άμεσα μόνο εσάς. Σήμερα δηλαδή συζητάμε με πέντε ή ε, έχουμε πέντε υποψήφιους ε, Μισό λεπτό διακόπτη πρόεδρος. Η επόμενη υποψήφια από το Λουξεμβούργο είναι μία κυρία. Α, τότε λέει ο μιλητής, ε, είχα λάθος ε, πληροφορίες. Ε, βλέπω όμως να υπάρχει μία ουσιαστική ανισορροπία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Δεν διαφυλάστε την αρχή της ισότητας των δύο φύλων. Ε, και μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Also ich glaube, dass das nicht ganz einfach ist für einen Kandidaten, sein eigenes Geschlecht in Frage zu stellen. Ich... Ε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική ως πρόεδρος, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά ξέρετε, θέλω να σας πω το εξή ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την υποβάλουμε στις κυβερνήσει. γιατί εδώ έχουμε έναν πολύ καλό υποψήφιο. Και τι να πει και εκείνο για αυτό το θέμα, δύσκολο να απαντήσει, αλλά, με πάση περιπτώσει, αν θέλει να απαντήσει, παρακαλώ, απαντήστε. Ε, ε, ε, νομίζω ότι, όπως λέει και η Πρόεδρος, εγώ δεν έχω κανένα ιδιαίτερο λόγο ή καμία ιδιότητα για να αποφανθώ για αυτό το θέμα. Ε, πολύ συχνά ήμουν υποψήφιος σε θέσεις που είχε και γυναίκες υποψήφιες και πήραν τις γυναίκες. Ε, τώρα ελπίζω να δεχτείτε μένα. Ε, εξ όσων γνωρίζω, και σας αποκαλύπτω και ένα μυστικό τώρα, υπήρχαν και άλλες υποψήφιες μάλλον άλλοι υποψήφοι για τη θέση αυτή, οι Γάλλοι, ε, χωρίς γυναίκα, καμία. Δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη επιλογή. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν έχει κανένα λόγο ε, στον ορισμό των υποψηφίων. Ε, και εύκολα εξηγείται αυτό. Και, και εξ όσου γνωρίζω, επίσης δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών για την επιλογή των υποψηφίων. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει αυτό και όσο δεν υπάρχει, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ισομερή εκπροσώπηση ή τουλάχιστον να την προσεγγίσουμε. Αυτά έχω να πω. Και σας ζητώ συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Ε, τι φταίτε εσείς, δεν, δεν φταίτε εσείς αλλά εμείς έχουμε μπροστά μας έναν πραγματικά ιδιαίτερα ικανό υποψήφιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε με τόσες πολλές λεπτομέρειες στις ερωτήσεις. Και τώρα, διακόπτη πρόεδρος. So, nun erwarten wir die Kandidatin. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε την κυρία υποψήφιο, υποψήφια για τη θέση επίση του ελεγκτή ελεκτικού συνεδρίου. Κυρία Ζωέλ Έλβιγκερ, παρακαλώ. Ich darf Sie ganz herzlich σας ε, καλωσορίζω θερμά, πολύ θερμά και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Κρέτην ο οποίος ε, ήρθε ε, την Ηλιάνα Ιβάνοβα. Επίσης, σας χαιρετίζω όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε και οι δυο σας εδώ σήμερα και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην κυρία Ελβίνκερ, αλλά πρώτα απ' όλα να παρουσιάσω τον εισηγητή ε, για την κυρία Ελβίνκερ, ο οποίος είναι ο κύριος Ολιβιέ Σαστέλ. Είναι ο εισηγητής ε, για την υποψηφιότητά της. Ε, και βεβαίως θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ελβίνκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, το πρώτο είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το γεγονός ότι μου δώσετε την ευκαιρία σήμερα να συστηθώ. Είμαι πεπισμένη Ευρωπαία και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα ε, να εκπροσωπώ το Λουξεμβούργο ως υποψήφια του Ελληνικού Συνεδρίου, να έρθω σήμερα εδώ και κυρίως να απαντήσω στις ερωτήσεις Όπως μπορείτε να δείτε από το βιογραφικό μου. Στη, μέχρι τώρα στα διοδρομία μου έχω συγκεντρώσει εμπειρία κυρίως για νομικά θέματα, ε, για το φορολογικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το εργασιακό δίκαιο. Ε, ως ε, πολιτική, ε, πολιτικός από το 2013 βουλευτής στο Λουξεμβούργο και ως δημοτικός σύμβουλος εδώ και αρκετά χρόνια επίσης μπόρεσα να συγκεντρώσω πολλές γνώσεις στους τομείς των δημόσιων οικονομικών, των φορολογικών και επίσης και της συνεργασία των θεσμών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε υψηλότερο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι με αυτές τις γνώσεις που έχω συγκεντρώσει και με την ε, εργασία μου θα μπορέσω και εγώ να προσφέρω κάτι στην εργασία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως νομικός τώρα στα γαλλικά έχω την απαραίτητη εμπειρία για την ανάλυση νομιμότητας και συμβατότητας με τους νόμους και τους κανονισμούς. Ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και του Προπολογισμού της Βουλής του Λουξεμβούργου εδώ και έξι χρόνια. Είχα την τιμή να διατελέσω εισηγήτρια της φορολογικής μεταρρύθμισης το 2016 και του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018. Εκτός από την εμπειρία μου, ε, ως προς την κατάρτιση και εκτέλεξη του προϋπολογισμού, αυτές οι δύο θέσεις που είχα ως εισηγήτρια μου επέτρεψαν να έχω βαθιά γνώση των δημοσίων οικονομικών ως αντιδήμαρχος αλλά και δήμαρχος στη συνέχεια ε, μπόρεσα να αποδείξω ότι ε, έχω ισχυρές ηγετικές και διαχειριστικές ικανότητες και ότι είμαι αφοσιωμένη στη φιδωλή, αποτελεσματική και αποδοτική ε, εκτέλεση των οικονομικών πόρων και στην προστασία των συμφερόντων των πολιτών. Στα αγγλικά τώρα η αγαστή συνεργασία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο είναι υψή τη σημασίας έτσι ώστε να σφυριλατηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν με επιβεβαιώσετε ως μέλος ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου θα κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώσω έτσι περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Οι καλές σχέσεις για μένα είναι ε, με βάση συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοώ και να λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ ταυτόχρονα θα σέβομαι και την αρχή της ανεξαρτησίας. Για το λόγο αυτό θα είμαι στη διάθεση του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της δικής σας Επιτροπής Ελέγχου του Περιπολογισμού για να είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο ε, να σας υποστηρίζω συζητώντας όποιο θέμα ενδιαφέρει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που με ε, ορίσετε μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, θα είμαι απολύτως ανεξάρτητη στην εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία θα εκτελώ πάντα προς το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύομαι ότι είμαι ανεξάρτητη και να είμαι ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό κόμμα και θα παραιτηθώ από οποιαδήποτε θέση κατέχω σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ε, θα κάνω τα καθήκοντά μου με ανεξαρτησία και αραιότητα, αμεροληψία και επαγγελματικό ε, ε, πνεύμα. Και ελπίζω να συνεισφέρω όσο μπορώ περισσότερες εργασίες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα σεβαστώ απολύτω το κώδικα δεοντολογίας και ηθική συμπεριφορά και πάντα ε, θα εργάζομαι προ το καλύτερο συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, ελπίζω να κερδίσω την εμπιστοσύνη σας και ε, να με ορίσετε μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Σα σας ευχαριστώ για την προσοχή σα και περιμένω με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ολιβιέ Σαστέλ, παρακαλώ να κάνει τι ερωτήσει του. Κυρία Έλβιγκερ, σας ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσίασή σας και για τις παρατηρήσεις, της γραπτές, τις οποίες στείλατε στα μέλη της Επιτροπής μας. Γνωρίζετε κι εσείς πως πέραν του δημοσιονομικού ελέγχου και των ελεγκτικών καθηκόντων θα πρέπει το ελεγκτικό συνέδριο να εστιάζει και στην απόδοση έτσι ώστε κάθε ευρώ να ε, επενδύεται και να δαπανάται με ευφυή τρόπο. Περιμένουν αυτό από εμά οι συμπολίτε μας, δεν υπάρχει πλέον τέτοιο θέμα. Πώς φαντάζεστε εσείς αυτούς τους δείκτες απόδοσης και πώς θα τους εντάξετε στον τρόπο με τον οποίο, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο θα σας ποιο χώρο θα αναλάβετε στο ελληνικό συνέδριο, πώς θα το κάνετε λοιπόν αυτό. Δεύτερον, εναρμόνιση των ελεγκτικών συστημάτων. Σύμφωνα με εσά και των γνώσεών σας, τα συστήματα αυτά δεν είναι πάντοτε εναρμονισμένα. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η εναρμόνιση, έτσι ώστε να είναι ε, μεγαλύτερος βαθμός αυτής από ό,τι σήμερα. Τρίτον, για την ε, διοικητική απλούστευση που χρειάζεται, γιατί όλα είναι περίπλοκα και δημιουργούνται σφάλματα. Τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να βελτιώσετε ε, αυτή την προσπάθεια για την διαχειριστική απλούστευση με τους εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, με τους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών και ποια είναι η σύνδεση των αποστολών μεταξύ ε, ε, της, του Ενακτικού Συνεδρίου, της Όλαφ και της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που σε λίγο θα ξεκινήσει να ε, λειτουργεί. Ποιος, πώς ε, συνδέονται οι, τα καθήκοντά σας και η αποστολή όλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σίγητα, για τις ερωτήσεις που κάνετε, για την πρώτη να σας πω πως για τους δείκτες απόδοσης είναι πολύ σημαντική για την ορθή ε, δημοσιονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων. Οι στόχοι που έχουμε θέσει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και επιτεύξιμοι. Εάν δεν είναι σαφείς, αν οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι περίπλοκοι, αν οι κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι σαφής τότε θα πρέπει εμείς να τους βελτιώσουμε με δείκτες απόδοσης, οι οποίοι θα ε, κάνουν τη μέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων και των ε, δημοσιονομικών επιπτώσεων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει όταν επιλέξουμε αυτούς τους δείκτες να το κάνουμε με προσοχή έτσι ώστε να δίνουμε τρίσιμα αποτελέσματα ε, για να γνωρίζουμε και τι πετύχαμε, αλλά και σε τι βαθμό το πετύχαμε. Ε, για την εναρμόνιση, να σας πω πως το ελεγκτικό συνέδριο ακολουθεί τους λογιστικούς κανόνες ε, που χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Είναι τα διεθνή πρότυπα in to και νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα κράτη-μέλη να έχουμε νομοθετικό υπερθεματισμό, έτσι ώστε οι οδηγίες οι οποίες εφαρμόζονται να είναι το κείμενο των οδηγιών, έτσι ώστε να μην έχουμε υπερβολική ρύθμιση η οποία θα έρχεται σε σύγκρουση με τα ε, ε, όσα επιδιώκουμε και με τους στόχους που έχουν θεσπίσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Euh, Οι ανταλλαγέ με τι αρμόδιε ελεγκτικέ αρχέ σε εθνικό επίπεδο, η ψηφιοποίηση νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση εδώ. Και όπω είπα και στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσα, καλό θα ήταν να έχουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα κοινή για όλους που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εθνικό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για να ανταλλάσσουμε στοιχεία περί μεθοδολογίας, για τα αποτελέσματα ελέγχων και η ψηφιοποίηση αυτή θα μας επιτρέψει να έχουμε τη βέλτιστη απόδοση των διαδικασιών ελέγχου και τα στοιχεία που έχουμε να είναι πιο καλά, πιο αξιόπιστα, πιο συγκεκριμένα, κάτι το οποίο θα είναι πλεονέκτημα ε, και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για την αποστολή του και τα καθήκοντα του ε, Ελεγκτικού Συνεδρίου και πώς συνδέονται με την Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Αγγελία, εμεί είμαστε ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι αποστολή μας ούτε να ανοιχνεύσουμε την απάτη και αν ανοιχνεύσουμε απάτη αμέσω τη στέλνουμε στην Όλαφ, η οποία ε, διώκει αυτές τις απάτες σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Συγγελία, η οποία θα ξεκινήσει το 2020 τη δράση της, θα παίξει ένα τεράστιο ρόλο στη μάχη για την καταστολή του διασυνοριακού εγκλήματος και κυρίως της απάτης, της διαφθοράς, και της επιβαρημένης ε, ε, απάτης στο χώρο του ΦΠΑ και θα αποφύγουμε έτσι ε, τη μακροχρονή διαδικασία δικαστικής συνδρομής, μια και πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της άριστης συνεργασίας αλλά και της αποδοτικής προσπάθειας έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Όλφ να συνεργαστούν με έναν τρόπο που με το βέλτιστο τρόπο θα πατάξει ε, το έγκλημα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριο Ζεντόφσκι παρακαλώ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κυρία Ελβίνγκερ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, βλέπω ότι όλοι λένε ότι χαιρόμαστε τελικά πάρα πολύ που προτείνονται και κάποιες γυναίκες για αυτή την τόσο σημαντική θέση. Εγώ δεν θα το παραλάβω βέβαια. Εγώ θα εστιάσω περισσότερο στο εξής. Τα μέσα ενημέρωση όταν ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά σας για αυτή την τόσο σημαντική θέση, ε, έγραψαν ε, για την οικογενειακή σας κατάσταση, και για τη σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει. Μήπως μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το δεύτερο ερώτημα, το δικό μου, αφορά στη δουλειά σας. Θέλουμε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς βλέπετε τη συνεργασία ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο και την Όλαφ και πώς ακριβώς Θεωρείτε ότι ε, πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία στο μέλλον ανάμεσα σε αυτούς τους τόσο δύο σημαντικούς ε, θεσμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα απαντήσω γαλλικά. Άρα, σε ό,τι αφορά την οικογενειακή μου κατάσταση, είναι γεγονός ότι ο πατέρας μου είναι ιδιοκτήτης ενός βιομηχανικού ομίλου Ωστόσο, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι προς το παρόν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας, ε, θέση από την οποία σκοπεύω να παρετηθώ. Οπωσδήποτε, σε περίπτωση που με ορίσετε μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Αλλιώς, ποτέ δεν συμμετείχα στην καθημερινή διοίκηση της επιχείρησης, ούτε κατέχω μετοχές στην εταιρεία είναι του πατέρα μου. Και σε ό,τι φορά μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, στο Λουξεμβουργό στη Βουλή δεν είχα ποτέ σύγκρουση συμφερόντων. Πάντα τηρούσα τον κώδικα δεντρολογίας και τον εσωτερικό κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων ε, στο Λουξεμβούργο. Το ίδιο θα πράξω ε, σε περίπτωση που με ορίστε μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα σέβομαι τον κώδικα και σε περίπτωση που ε, υπάρξει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων θα ενημερώσω τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου και θα ζητήσω ε, από τον πρόεδρο να μην είμαι μέλος του δεύτερου τμήματος έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία ε, ελεκτικού συνεδρίου και Όλαφ. Τη υπηρεσία ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αρμόδια για την απάτη και την καταπολέμησή τη. Ε, νομίζω ότι είναι εκ των όνων κάνευ αυτή η συνεργασία για να καταπολεμάται η απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα και ο προπολογισμό της Ένωσης από απάτες, οργανωμένο έγκλημα και οποιαδήποτε διαφθορά. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει ως αποστολή την ανείχνευση ε, απάτης, αλλά σε περίπτωση που υποπτεύεται τέτοια ε, απάτη, τη βρίσκει σε έλεγχο, είναι υποχρεωμένο το ελεγκτικό συνέδριο να τα διαβιβάζει στην Όλαφ. Δεν έχει ούτε ανακριτικές αρμοδιότητες, ερευνητικές, ούτε ε, πειθαρχικές επιβολής κυρώσεων. Οπότε εγώ προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή τη συνεργασία σε περίπτωση που με ορίσετε, Ενδεχομένω να δούμε εσωτερικά στο ελεγκτικό συνέδριο που μπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Ε, ε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επόμενη ερωτώσα, Λάρα Βόλτερς, από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Η ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά ε, στις απάτες, στις φορολογικές και στη φοροδιαφυγή. Από τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις μάλλον που μας έχετε στείλει σε γραπτή μορφή, γνωρίζω ότι έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα και μπορώ να φανταστώ ότι ίσως να μην ασχοληθείτε με το θέμα αυτό στο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και η δική μου ερώτηση είναι, μετά τα Panama Papers, τα LuxLeaks και τα συναφή, θεωρείτε εσείς ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο ε, πώς βλέπετε ακριβώς το να εξελίσσεται ο ρόλος του ελληνικού συνεδρίου σε αυτό τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, νομίζω ότι το τμήμα υπαριθμών 4 είναι εκείνο το οποίο ασχολείται με το θέμα έχω δει ότι έχει γίνει εκεί ένας έλεγχος και υπάρχει και μία έκθεση η οποία βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος που διαδραματίζει το ελεγκτικό συνέδριο είναι σημαντικός όσον αφορά στη φοροδιαφυγή. Γενικά, εγώ έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα ε, στο Λουξεμβούργο και το Λουξεμβούργο έχει υιοθετήσει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες ε, επί του θέματος ε, το έγγραφο 5, το 6, τώρα πρόκειται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο καλείται να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα, σε αυτόν τον τομέα και νομίζω ότι η ψηφιοποίηση ε, θα είναι πρόκληση για το ελεγκτικό συνέδριο. Γιατί όσο περισσότερο θα ψηφιοποιούνται τα αποτελέσματα σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ανώτατων θεσμών των κρατών μελών, αυτό θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μας να κάνουμε καλύτερους ελέγχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Πέξα. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που υπάρχει να συζητήσουμε μαζί σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ, πολύ ωραία αυτή η έκπλαξη. Ε, μία μικρή χώρα, όπως είναι το Λουξεμβούργο, να φροντίζει για την ισότητα των δύο φίλων στο ελεγκτικό συνέδριο. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά επίσης τη φοροδιαφυγή. Στις ε, γραπτές ερωτήσεις απαντήσατε ότι ως μέλος του Κοινοβουλίου είχα την ευκαιρία να ελέγξω ουσιαστικά το τι έκανε το Λουξεμβούργο για να εφαρμόζει τις ε, διατάξεις και τις ε, νομοθεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις, τους, ευρω... τους διεθνείς κανονισμούς. Έχουν γίνει κάποιες νομοθετικές αλλαγές αλλά παρόλα αυτά το Λουξεμβούργο εξακολουθεί να θεωρείται φορολογικό φορολογικός ε, παράδεισος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι η ε, πολιτική ομάδα ε, στην οποία ανήκει ο βουλευτής από το χώρα σας είναι υπέρ του κράτους δικαίου με μία εξαίρεση όταν ο κύριος Μπάμπης βρέθηκε σε σύγκρουση συμφερόντων δηλαδή πήρε χρήματα από το ε, ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό και παράλληλα ήταν εκείνος που έπρεπε να αποφασίσει πού θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, σε περιπτώσεις όπου η χρήση κονδυλίων ελέγχεται σε κράτη-μέλη η Renew Europe όπου βρίσκεται στην κυβέρνηση. Τι ακριβώ πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει για αυτέ τέτοιου είδου περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας. Η πρώτη ερώτηση αφορά στη φοροδιαφυγή και την ε, κατάσταση στο Λουξεμβούργο μετά τα LuxLeaks. Το Λουξεμβούργο από το 2013 έχει καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες να συμμορφωθεί πλήρως ε, και το Φόρουμ Μοντιάλ για τη Διαφάνεια. Επίσης, ε, έχει ταξινομήσει το Λουξεμβούργο σε μια χώρα που έχει συμμορφωθεί απόλυτα. Το Λουξεμβούργο έχει ε, υπογράψει πάρα πολλές ε, συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης, ε, ε, νομίζω πάνω από 80, με 80 χώρες του κόσμου. Έχουμε εφαρμόσει την οδηγία DOC5, την MID. Επίσης, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει ή μάλλον έχουμε καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες όσον αφορά τη διαφάνεια τα τελευταία 6 χρόνια. Η ΦΑΤΚΑ, η συμφωνία το 2014 υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων έχουμε επίσης ε, διευρύνει ε, την ε, αντιμετώπιση του ε, ξεπλήματος ε, χρήματος την έχουμε αναγάγει σε ποινικό αδίκημα, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες και από τις συστάσεις από το 12 μέχρι το 14. Η DOC 6, όπως σας είπα, βρίσκεται στη φάση όπου πρόκειται να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο να θεσπιστεί και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τον προεπολογισμό του 2020, ο Πεκαμίνιο, ο υπουργό μας των Οικονομικών, ανακοίνωσε επίσης ότι όλες οι συμφωνίες υφαλογικές που είχαν ε, θεσπιστεί πριν από τον Ιανουάριο του 2015 δεν θα ισχύουν πλέον μετά τον Ιανουάριο του 2020, αλλά δηλαδή όλες οι προγενέστερες συμφωνίες ε, θα περιορίζονται σε μια διάρκεια ισχύω 5 ετών. Ε, δεν ξέρω. τι ήταν ίσως ε, η ερώτηση για την ερώτησή σας. Εγώ ε, δεν θεωρώ ότι το Λουξεμβούργο μπορεί να συγκριθεί με τα νησιά Καϊμάν, παραδείγματος χάρη. Και αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς δεν ξέρω αν με αφορούν, γιατί αφορούν την περίοδο πριν εγώ ασχοληθώ με την πολιτική και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες σε αυτό τον τομέα. Όσον αφορά στην ανεξαρτησία του συνεδρίου όταν γίνονται έλεγχοι στα κράτη-μέλη, εγώ βεβαίως ε, το δικό, μου, το δικό μου το κράτος ε, το βάζω στην ίδια μοίρα όπως και όλα τα άλλα κράτη και θα κάνω την, τους ελέγχους ε, με πλήρη ανεξαρτησία είτε πρόκειται για έλεγχο σε Λουξεμβρούγο είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Άλλη μια ερώτηση από τον κύριο Αντινόλφη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την ε, εισήγηση της υποψηφίου και πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την υποτιθέμενη ανεξαρτησία ε, από την μεγάλη αυτή εταιρεία, τον όμιλο επιχειρήσεων που κατέχει η οικογένειά της. Στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις, ε, μέλη οικογένεια αποφεύγουν να ενταχθούν σε μεγάλους θεσμούς και οργανισμούς. Γιατί, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο ε, νομίζω ότι είναι ε, προσβολή της ευφύειας. Το Λουξεμβούργο εδώ και πέντε χρόνια ε, συμμετέχει στη φορολογία των εξωτερικών επιχειρήσεων και είναι γνωστό ότι το Λουξεμβούργο νομίζω ότι έχει βρεθεί σε μια θέση όπου αντιμετωπίζει αθέμητο ανταγωνισμό, κατηγορίες για αθέμητο ανταγωνισμό από άλλα κράτη-μέλη. Αλλά δηλαδή αυτά ε, οι διαβεβαιώσει εκ μέρου του Λουξεμβούργου πραγματικά θεωρώ ότι είναι προσβολή στην ευφυΐα όλων των κρατών μελών, ε, έναντι όλων των χωρών που βρέθηκαν σε κρίση όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι αυτά είναι προσβολή οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν κρίσεις και το Λουξεμβούργο εδώ και χρόνια εφαρμόζει μια φορολογία σκανδαλώδη έναντι των πολυεθνικών. Έχει γίνει ε, κάποια, ε, θεωρώ μάλλον, ή περισσότερο να ρωτήσω, ε, πιστεύετε ότι πρέπει να αναλυφθούν κάποιες ενέργειες για να αποφευθεί αυτή η στάση που κρατάει το Λουξεμβούργο έναντι των πολυεθνικών εταιριών. Θα ήθελα να πω στους ερωτώντες, ε, κοιτάξτε, αν υπάρχουν ε, ερωτήσεις, που έχετε να κάνετε, μην ξεχνάτε ότι όταν πρόκειται για εθνικές αποφάσεις, τι να κάνουν και τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Δεν μπορούμε και να στιγματίσουμε και κανέναν ε, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Εμείς είμαστε εδώ για την στάση του καθενός μεμονωμένου υποψηφίου. Τα λέω αυτά έτσι πολύ προσεκτικά, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λιγάκι δίκαιοι έναντι των υποψηφίων και να παραμένουμε και αμερόληπτοι ή δυνατόν. Euh, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς για τις ερωτήσεις σας. Για την οικογενειακή επιχείρηση, όπως σας είπα, προσωπικά δεν έχω μετοχές στην εταιρεία. Δεν είχα ποτέ. Άρα λοιπόν δεν βλέπω γιατί προσωπικά τώρα έχω σύγκρουση συμφερόντων. Όπως σας είπα, θα ζητήσω ε, να μην είμαι παράλληλα πρόεδρος του δεύτερου τμήματος. Είναι όμως εταιρεία του πατέρα μου και δεν μπορώ να του ζητήσω να την πουλήσει αύριο γιατί εγώ έκανα την συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή προσωπικά. Θα μπορούσα να έχω ε, δουλέψει και εγώ στην οικογενειακή επιχείρηση επιλογή μου ήταν να ανεξαρτοποιηθώ, να γίνω δικηγόρος και να κάνω πολιτική καριέρα κατόπιν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποφύγω οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την οικογενειακή επιχείρηση στην οποία δεν εργάστηκα ποτέ. Τουλάχιστον δεν μισθοδοτήθηκα ποτέ. για τα φορολογικά θέματα του Λουξεμβούργου. Δεν θεωρώ ότι βλάπτει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και όπως απάντησα στα... στη συνάδελφό σας κυρία Βάουτερς και στον κύριο Πέξα, το Λουξεμβούργο ε, αξιολογήθηκε και θεωρήθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια ως σε μεγάλο βαθμό σύμμορφο, largely compliant. Δεν είμαστε σε κανένα κατάλογο, μαύρο κατάλογο. Έχουμε μεταφέρει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως θα έπρεπε μέχρι σήμερα. Δεν θα ήθελα εδώ να ακούσω πως εμείς ε, φορολογούμε με έναν τρόπο που βλάπτει το υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είμαστε ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα αφοσιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυβερνητική εταίροι όπως και η κυβέρνηση πρώτου 2013, έχουν πάντα υποστηρίξει τη διαφάνεια και πάντα εργαστεί υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λιγάκι για να χαμογελάσετε και λίγο. Αυτή η συνεργασία είχε ε, μια πολύ καλή και μακρά συνεργασία με τον συνάδελφό σα από το Λουξεμβούργο. Γνωρίζει την Επιτροπή, ε, γνωρίζει το Ελληνικό Συνέδριο. Από μέσα και απ' έξω, επιτρέψτε μου ε, μια πολύ προκλητική ερώτηση. Εσείς τι προτείνετε να κάνετε, νομίζετε ότι θα καταφέρετε να τα κάνετε καλύτερα από τον προκάτοχό σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ θα το κάνω. Αλλά θα είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο να ε, ανταγωνιστώ ε, την εμπειρία του προκατόχου μου, ο οποίος πραγματικά έκανε μια καταπληκτική δουλειά στο ελεγκτικό συνέδριο, αλλά θα κάνω, με πάση περιπτώσει, ό,τι μπορώ, έτσι ώστε να είμαι τουλάχιστον τόσο καλή και αυτός. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ε, νομίζω ότι τώρα πια δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen. Κάτι δεν κατάλαβα καλά. Νομίζω ότι κανονικά θα είχαμε λίγο χρόνο, αλλά ήρθε και ο πρόεδρος λίγο νωρίτερα, οπότε πάει και ο χρόνος. Alles gut. Wir hätten dich ja vorher reingelassen. Okay. So, ich begrüße Καλωσορίζω θερμότατα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και χαίρομαι ε, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την ακρόασή του ε, για το νέο του διορισμό. Έχουμε μισή ώρα. Εισηγητής μας είναι ο κύριος Στεχόφσκι. Έχουμε κάνει ήδη τρεις ακροάσεις σήμερα. Η τέταρτη είναι τούτη εδώ. Και Παρακαλώ τον κύριο Λένε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Λοιπόν, εδώ και έξι χρόνια έχω την τιμή και το προνόμιο να προείσταμαι ενός ε, θεσμού που έχει ένα ιδιαίτερο καθήκον. Ειδικά σήμερα στους ε, ταραγμένους καιρούς, ε, το ελεγκτικό συνέδριο ως ελεγκτής των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πολύ σημαντικός. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ηττίας μου νομίζω ότι απέδειξα ότι έχω συμβάλει και εγώ στην τόσο σημαντική εργασία του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό, κατά την άποψή μου, φαίνεται και το γεγονός ότι οι συνάδελφοι από το ελεκτικό συνέδριο εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου για μια δεύτερη θητεία. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν χρόνια επιτυχίας για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Μπορέσαμε να καταρτήσουμε μια ε, στρατηγική που είναι στραμμένη προς το μέλλον και να την εφαρμόσουμε. Το 2016 όταν υπέβαλα υποψηφιότητα είχα πει ότι το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να αποδείξει θέμενη αξία όσον αφορά τι αιτήσει εκθέσει, τι δηλώσει αξιοπιστίας, να εστιάσει την προσοχή του σε πολλά και διαφορετικά οικονομικά θέματα. Τους στόχους αυτούς ε, για το 2018 έω 2020 τους ε, θέσαμε και πάλι στον εαυτό μας και έκτοτε νομίζω ότι έχουμε επιτύχει αρκετά σημαντική πρόοδο. Το ελεγκτικό συνέδριο όλο και περισσότερο συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων στη δουλειά του, Κάνουμε πολλούς σημαντικούς ελέγχους, ε, βεβαίως χωρίς να παραμελούμε τη συμμόρφωση. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο είναι εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών και ενδιαφέρεται και κατά πόσο παραδείγματο χάρη το αεροδρόμιο που έχει κατασκευαστεί είχε νόημα, κατά πόσον χρησιμοποιείται και κατά πόσον αυτό έχει εξίσου νόημα όπως ε, και στους, το αν στους κανονισμούς, στους διαγωνισμούς που προκυρήσονται τηρούνται όλες οι προδιαγραφές. Τα τελευταία χρόνια ε, συνεργαζόμαστε πιο πολύ με εκείνους ε, που, στους οποίους απευθυνόμαστε και με άλλους ελεγκτικούς οργανισμούς. Σήμερα λοιπόν είμαστε περισσότερο ε, παρόντες στους stakeholders μας και κυρίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μένα πάντα ήταν πολύ σημαντικό η εμβάθυνση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και κυρίως με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Νομίζω ότι η προοπτική για μένα, επειδή ήμουν παλαιότερα νωρίτερα ε, Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το γεγονό ότι ήμουν ευρωβουλευτής. Ε, θεωρώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο προσφέρει υπηρεσίε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκθέσει μας έχουν ω νόημα να βοηθούν τον έλεγχο και να βελτιώνεται η νομοθεσία. Αυτό πάλι προποθέτει ότι τα θέματα που είναι σημαντικά για εσά πρέπει να τα εξετάζουμε και να σας παρουσιάζουμε έγκαιρα τα συμπεράσματά μα. Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού. Βελτιώσαμε τον προγραμματισμό με περισσότερο ε, στρατηγική κατεύθυνση. Τώρα λοιπόν εξετάζουμε αυτά που μας προτείνεται, τα εντάσσουμε στη δουλειά μας και έτσι οι μισές από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται πλέον ε, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας μας. Εάν λοιπόν ε, ανανεώσετε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, τότε και εγώ θα προσπαθήσω ακόμα περισσότερο να καταστήσω το ελεγκτικό συνέδριο πιο αποτελεσματικό και σημαντικό για για για την καθημερινή σας δουλειά. Πρόσφατα συστήσαμε ε, μία ομάδα εργασία με τον τίτλο Future Foresight, η οποία ομάδα εργασία ε, θα εργαστεί για την επεξεργασία της στρατηγικής μας για τα επόμενα χρόνια. Και εγώ θα μεριμνήσω έτσι ώστε τον δρόμο που έχουμε χαράξει να τον εκμεταλλευτούμε, να ε, εστιάσουμε περισσότερο σε ελέγχους και σε καλύτερη συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επίσης, με ενδιαφέρει η περαιτέρω βελτιστοποίηση του εσωτερική της εσωτερικής μας οργάνωσης για το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Θα δουλέψουμε. Πρώτο βήμα, ε, κατά την άποψή μου, έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, έχουμε βάλει ως στόχος ε, το ποσοστό των γυναικών στη διαχείριση μέσω πρόθεσμα να αυξηθεί στο 40%. Όταν εμεί ξεκινήσαμε πριν από 6 χρόνια, τότε ε, στο ελεγκτικό συνέδριο είχαμε μόνο δύο γυναίκες διευθύντρες και όταν επρόκειτο για το θέμα της προαγωγής υπήρχε το πρόβλημα ότι στη μεσαία βαθμίδα δεν υπήρχε σχεδόν καμία γυναίκα. Νομίζω λοιπόν τα τελευταία 6 χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Σήμερα έχουμε πολλά ε, καλά στελέχη γυναίκες οι οποίες είναι πολύ καλές για το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, και τέλος, όπως και μέχρι τώρα, θα θελήσω να έχω πολύ καλή σχέση με την Επιτροπή σας. Ε, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Το ελεγκτικό συνέδριο τίνει ευήκον ους ε, για τις προτάσεις που έρχονται από τη δική σας αλλά και από άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και βεβαίως και εμείς στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ο εισηγητής κύριος Ντεχόφσκι έχει το λόγο. Ε, οκ, okay, κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις έχω να σας κάνω η Μαρτίνα έκλεισε την περασμένη συζήτηση με μια πολύ προβοκατόρικη ερώτηση και θέλω και εγώ να σας προβοκάρω. Γιατί ξανακατεβαίνετε υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολύ επιτυχημένη. Τώρα δεν θέλετε να ξεχουραστείτε και να κάνετε κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι τα τρία σημεία που σας κάνουν να νιώθετε αυτή την ανάγκη να συνεχίσετε σε αυτή τη θέση. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την απόδοση και εστιάζω το εξής. Πώς θα βελτιώσετε τη δουλειά σας. Πώς θα παρουσιάσετε καλύτερα τις εκθέσεις σας στον κόσμο. Πώς θα δείξετε ότι είστε πολύ ισχυρός οργανισμός με απόλυτη διαφάνεια όσο και ανεξαρτησία. Και η τρίτη ερώτηση αφορά τη μελλοντική σας συνεργασία με την Όλαφ. Πολλοί από εμά γνωρίζουμε ότι κάνατε καταπληκτική δουλειά στη διερεύνηση της υπόθεσης του ΕΑΖΟ, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου, σε στενή συνεργασία με την Όλαφ. Τώρα συζητούμε το θέμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και η Όλαφ θα γνωρίσει περικοπές στο προσωπικό της. Στο μέλλον, πώς ε, προβλέπει; Ναι, ναι, τους κόβουμε 80 άτομα από την Όλαφ ε, για το μέλλον, γιατί τους θέλουμε στην εισαγγελία να εργαστούν. 50 με 80 είναι περίπου οι περικοπές ε, των θέσεων. Ε, άρα στο μέλλον χρειάζεται ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών ε, εξαρτήτων θεσμών. Ξέρω ότι εσείς έχετε διακριτό ρόλο. Η Όλαφ ε, κάνει τις ανακρίσεις και τις έρευνες και εσείς το λογιστικό έλεγχο. Όταν το συζητήσαμε αυτό με το διευθυντή της Όλαφ, μας είπε ότι εκτιμάει πάρα πολύ τη συνεργασία και την κατάρτιση. Πολύ σύντομα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Ja, Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, κύριε Βουλευτά. Κοιτάξτε το γιατί που ρωτήσατε, ε, πολύ απλή αράτηση. Πρώτον, γιατί μου κάνει κέφι. Κοιτάξτε, μου κάνει κέφι, το, το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι ότι φέτος έγινε 62 χρονών δεν είμαι παλιοκαραβάνα, δεν γέρασα, αλλά έξι χρόνια μπορώ μια χαρά να δουλέψω. Και δεν θέλω να βγω σε πρόορη σύνταξη. Ο τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα έξι χρόνια έμαθα ότι πράγμα, πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν και στο ελεγκτικό συνέδριο και εκτός αυτού. Γιατί το ελεγκτικό συνέδριο, λόγω του γεγονότος ότι είναι ανεξάρτητος οργανισμός, ότι έχει πάρα πολλούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, έχει πολύ καλή φήμη. Και όταν λέει κάτι το ελεγκτικό συνέδριο, αυτό έχει βαρύτητα. Και το να ε, εκφράζει κανείς το ελεγκτικό συνέδριο προς τα έξω και να προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα, έστω και έμεσα, μέσα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ε, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε, αυτό δίνει σε κάποιον το αίσθημα της επιτυχίας. Και αυτοί είναι οι τρεις λόγοι, γιατί είπα και εγώ, ναι, εγώ θα ήθελα να δουλέψω άλλα έξι χρόνια. Στο ερώτημα τι μπορούμε να βελτιώσουμε, καταρχήν θέλω να πω ότι ε, τα τελευταία τρία χρόνια ε, της Προεδρίας μου και τα έξι γενικότερα καταφέραμε πάρα πολλά. Δηλαδή ε, διπλασιάσαμε τις πληροφορίες που δίνουμε στα μέσα ενημέρωσης. Επίσης, εκτός από τις αιτήσεις εκθέσεις, διπλασιάσαμε πολλά άλλα που δίνουμε προς τα έξω. Τις επαφές με τους stakeholders ε, και αυτές τις εντατικοποίησαμε. Και εντάξει, δεν είναι δικό μου επίτευγμα αυτό, είναι επίτευγμα μιας ολόκληρης ομάδας. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις και τώρα έχουμε μια ενδιάμεση έκθεση για το peer review που ανατέσαμε ε, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής μας. Και η peer review, ε, όσοι ασχολήθηκαν με αυτό, ε, ήταν πολύ επιφυλακτική, είδαν τους στόχους της στρατηγικής, είδαν τι έχει επιτευχθεί τα πρώτα τρία χρόνια και ξέρετε κάτι, υπάρχουν τομείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. Παραδείγματο χάρη, μεταρρύθμιση της ετήσιας έκθεσης. Εκεί πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι έλεγχος που βασίζεται περισσότερο σε συμπεράσματα άλλων ελέγχων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε. Άρα δηλαδή όλα αυτά ε, συνδέονται έμεσα και με το πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε κονδύλια για περαιτέρω δραστηριότητες ε, που να έχουν αποτέλεσμα. Ως ε, ελεγκτικό συνέδριο στην διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών που έχω την τιμή να εμφανίζω μια φορά το χρόνο από την διάσκεψη των Προέδρων αυτών παίρνουμε κάθε χρόνο 60 προτάσεις για τις εκθέσεις αυτό λοιπόν δείχνει ότι προφανώς ε, η ζήτηση ε, για την απόδοση για performance είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά και εγώ αυτά μπορώ να τα πετύχω μόνο αν έχω τα κονδύλια να τα χρησιμοποιώ πιο αποτελεσματικά για να πετύχουμε το στόχο. Τώρα, όσον αφορά την σπουδαιότητα ε, των εκθέσεων, αυτό το Future Foresight παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν άλλα ελεκτικά συνέδρια, το Αμερικανικό, οι Φινλανδοί συναδελφοί, ότι αυτοί τα καταφέρνουν, ε, έχουν μικρές μονάδες οι οποίες ε, δικτυώνονται με άλλους θεσμούς ε, που υπάρχουν στην Ευρώπη και ασχολούνται με το Future Foresight. Και τι γίνεται. Ε, παίρνουν ερωτήσεις και ιδέες από όλους αυτούς και μετά ελέγχουν κατά πόσον αυτά μπορούν να παίξουν ρόλο για μελλοντικούς ελέγχους. Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν κρίσεις ε, που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Είναι και αδύνατον. Όπως ας πούμε στην οικονομική κρίση του 2008 ήταν αδύνατον και δεν μπορεί κανείς να προετοιμαστεί. Όμως υπάρχουν άλλες εξελίξεις για τις οποίες μπορούμε να προετοιμαστούμε. Πριν από δύο-τρία χρόνια συζητήσαμε στο συνέδριο ε, για το κατά πόσον παραδείγματος χάρη είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν έλεγχο την κυβερνοασφάλεια. Και τότε κοιταχτήκαμε και είπαμε μπα, μάλλον δεν γίνεται. Όμως αυτή είναι μια εξέλιξη που μπορεί κανείς και πρέπει να προβλέψει και όπου πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε εφόσον προβλέπει να προσαρμοστεί και να είναι σε θέση να αντιδράσει. Ως εκ τούτου εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα, το θέμα της προβλεψιμότητας, ε, του προσανατολισμού σε νέα σημαντικά θέματα για τα οποία πρέπει πρέπει ήδη το να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε στρατηγική. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο από το 20 και μετά. Ο κύριος Φιγκουρέντο είναι ο επικεφαλής αυτής της ομάδας εργασίας και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταθέσει σημαντικές προτάσεις στο ε, συνέδριο και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα εφαρμόσω. Για την Όλαφ, είπατε ότι μας είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς κάνουμε ελέγχους. Δηλαδή, εμείς δεν κάνουμε συγκεκριμένες έρευνες, ανακρίσεις για να αποκαλύψουμε απάτες. Ε, προσκρούμε κατά τύχει συνήθω σε απάτη, δηλαδή εξετάζουμε περιπτώσεις όπου βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες υπόνοιε. αυτές τις διαβάζουμε στην Όλαφ. Ας πούμε πριν από λίγους μήνες ε, ε, υπογράψαμε ένα, μια συμφωνία συνεργασία με την Όλαφ που προβλέπει ακριβώς αυτές τις διαδικασίε πώ θα αντιμετωπίζονται τέτοιου είδου περιπτώσεις και τι θα παραπέμπουμε εμείς ε, στην Όλαφ. Με το EPPO θα κάνουμε Ακριβώς το ίδιο. Ε, με την κυρία Βέζη, νομίζω λέγεται, ε, πρόεδρο της ΕΠΠΟ, ε, έγραψα, συνεργάστηκα μαζί της και είπε ότι μόλις αρχίσει να λειτουργεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ΕΠΠΟ, όπως την είπα, θα είμαστε σε πολύ πιο στενή συνεργασία. Θα έχουμε το τρίγωνο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ΕΚΟ και ελεκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Νομίζω αυτά ήταν τα τρία ερωτήματα που υποβάλλατε. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές και δημοκράτες, ε, συνάδελφος ε, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να κάνετε αυτή τη λεπτομερή ε, παρουσίαση και για τις απαντήσεις που θα μας δώσετε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε αρκετά ε, στην παρουσίαση που κάνατε ε, της ετήσιας έκθεσης, όπου αναφερθήκατε κάποιο πιλωτικό project μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και κρατών μελών τη στιγμή της προετοιμασίας των ελέγχων. Δώστε μας κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Δεύτερον, στη γραπτή σας απάντηση αναφέρεστε στην ανάγκη να ενισχυθεί η απόδοση και όχι τόσο πολύ η συμμόρφωση της μελλοντική σας εργασίας. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό δεν θα μειώσει τη συμμόρφωση, αλλά θα ήθελα να με εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Και τέλος, ένα θέμα που είχε εμφανιστεί στις ειδικέ εκθέσεις του Λεκτικού Συνεδρίου για τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν οι εθνικές αρχές σε κάποιους από τους κανόνες και κυρίως στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Φέτος, σε πέντε παρατηρήσεις αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, ε, παρατηρήσεις και συστάσεις δικές σας για τον τομέα της συνοχής όπου λέγεται πως οι εθνικές αρχές έχουν διαφορετική ερμηνεία στο πώς εφαρμόζονται και οι κανόνες. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσετε. Επίσης, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό στο μέλλον έτσι ώστε να μην ξαναεμφανιστεί. Ευχαριστώ. Επάντηση, ευχαριστώ πολύ. Για το πιλωτικό πρόγραμμα έχετε δίκιο ε, σε σχέση με τη μετάβαση, το λεγόμενο attestation audit, ε, στην ετήσια έκθεση για τη συνοχή αρχίσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο προσκρούει σε κάποια τεχνικά προβλήματα και αυτό το έχουμε δει. Για ποιο λόγο. Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη κάνουν το λογιστικό έλεγχο δεν ταυτίζεται με τη δική μας μεθοδολογία ούτε αντίληψη. Γι' αυτό υπάρχουν δυσκολίες ε, στην επαλήθευση των αποτελεσμάτων που μας έφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα το, ε, θέλαμε να το εντάξουμε στην ετήσια έκθεσή μας του χρόνου το 2020 θα κάνουμε μια ειδική έκθεση, την οποία πρόσφατα αποφασίσαμε στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας για το 2020 που θα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και αυτές τις δυσκολίες και θα το αναλύσει αυτό σε σχέση με το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα, θα το περιγράψει και μετά θα δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την παράλληλη ε, επιδίωξη συμμόρφωσης και απόδοσης απαντώ ως εξής. Στη δεκαετία του 90 θα θυμάστε όλοι φαντάζομαι ακόμα και όσοι δεν ήσασταν τότε βουλευτές έχετε διαβάσει εφημερίδες και ιστορία το 1999 ανάγκασε σε παρέτηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Επιτροπή Σαντέρ. Από το 1994 είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε βάσει της συνθήκη του Μαστρίχτ ε, δήλωση αξιοπιστίας στην ετήσια έκθεση. Από το 1994 μέχρι πριν από μία τριετία ε, κάθε χρόνο ήταν αρνητική η δήλωση αξιοπιστίας. Για ποιο λόγο. Τα σφάλματα ε, στη δεκαετία του 90 δεν τα δημοσιεύαμε, αλλά σε αποφασιστικούς τομείς ήταν διψήφια ε, οπότε, αν δούμε την κατάσταση τότε και τη συγκρίνουμε με τη σημερινή, η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει και δραματικά βελτιώθηκε, έστω και αν άργησε να πάρει μπρο μετά το 2001. Και αυτό πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να επιμείνουμε πάρα πολύ τώρα στη συμμόρφωση, γιατί έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία η απόδοση και επιδόσεις όχι μόνο για μας, αλλά και για τους εμπλεκομένους προφανέστατα. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο είναι. Αν συζητήσετε με τους προέδρους των επιτροπών, αυτό που τους ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι η απόδοση. Για να σας εξηγήσω. Ας πούμε, φτιάχνουμε ένα τερματικό σε ένα λιμάνι, σε ένα αεροδρόμιο ή σε μια γέφυρα. Αν πάει κάτι στραβά στην προκήρυξη, δεν μιλάω για απάτη ή διαφθορά, μπορεί να γίνει ένα λάθος, γιατί είναι περίπλοκοι οι κανόνες στην έγκριση του έργου. Μπορεί αυτό να δοθεί σε λάθος ανάδοχο. Αυτό είναι λάθος για τη συμμόρφωση, αλλά είναι λιγότερο σημαντικό από το να χτίσει το λιμάνι ή το αεροδρόμιο ε, ή αν έχει νόημα αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Χρησιμοποιούνται αυτά τα λιμάνια, υπάρχει ενδοχώρα, υπάρχουν δρόμοι που να φτάνουν εκεί στο αεροδρόμιο ή σε αυτό τον αυτοκινητόδρομο. Ε, είναι... Ε, μια δαπάνη ατελέσφορη ή συνδέεται με κάποιους συγκεκριμένους στόχους και πιάνει τόπο αυτή η επένδυση. Φυσικά δεν πρόκειται να παραμελήσουμε καθόλου τη συμμόρφωση με τους κανόνες, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι περισσότερο πια η απόδοση, αυτό το performance. Τώρα, τι κάνουμε όταν είναι διαφορετικές οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δεν είμαστε δικαστήριο υπό την έννοια αυτή. Εμείς βγάζουμε αποφάσεις, ε, εκδίδουμε συμπεράσματα, αλλά αυτά δεν είναι εκτελεστά. Μπορεί να διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν διαφωνεί, με της με χαρά της εάν συμφωνεί ε, μαζί μας, είναι ε, δικό της καθήκον ε, και καθήκον του Συμβουλίου να τα κοιτάξει αυτά και να την οθήσει προς την κατεύθυνση να αναθεωρήσει. Εμείς δεν μπορούμε να την αναγκάσουμε. Διάλογο κάνουμε και αυτό συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τις διαφορές της απόψης των κρατών μελών. Πολύ συχνά έρχομαι αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα. Από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη χώρα μου, βλέπω να έρχονται συχνά υψηλόβαθμα στελέχη ε, κυβερνήσεων κρατηδίων, πρωθυπουργοί κρατηδίων, υπουργοί οικονομικών ε, και οικονομίας και διαμαρτύρονται ότι το τοπικό τους ελεγκτικό συνέδριο έχει διαφορετική θεώρηση ε, και κάνει έναν έλεγχο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς όταν επισκεπτόμαστε εκεί. Και αυτό που τους λέω και τους προσφέρω είναι το εξής. Μπορείτε να μας ρωτάτε, δηλαδή και τα τοπικά ελεγκτικά συνέδρια, οι τοπικέ κυβερνήσει, εθνικέ κυβερνήσει. Δεν απαγορεύεται να μα στείλουν ένα γράμμα, να μα ρωτήσουν αυτό πώ το βλέπετε το θέμα. Και βεβαίω ε, εμεί γνωμοδοτούμε και με χαρά το κάνουμε. Βέβαια, εναπόκειται ε, στο, στο ελεγκτικό συνέδριο, τι τοπικές αρχέ ή τι εθνικές, να αξιολογήσουν την άποψή μας και να αποφασίσουν εκείνοι, γνωρίζοντας όμως τη δική μας άποψη. Εμείς δεν έχουμε ε, ε, μια δυνατότητα όπως έχουν τα δικαστήρια ε, να βγάζουμε μια απόφαση και να τη διαβιβάζουμε αρμοδίως ανωτέρως για να αποφασίσουν. Τη γνώμη μας λέμε. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το Ρινιού, Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που συμμεριστήκατε μαζί μας την ε, ανανεωμένη σας φιλοδοξία για το ελεκτικό συνέδριο. Θέλετε να είναι ακόμα ε, πιο αποδοτικό από ό,τι στο παρελθόν. Έχετε υπόψη ένα θέμα, ένα φάκελο που νομίζετε ότι το ελεκτικό συνέδριο θα μπορούσε να το έχει χειριστεί διαφορετικά ή καλύτερα για να εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο τον Ευρωπαίο πολίτη. Έχω και δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Δεν είναι πάρα πολύ ευρέω γνωστή η δουλειά που κάνει το ελεκτικό συνέδριο στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες στο ελεκτικό συνέδριο για να αποδείξει στους Ευρωπαίους πολίτες την προστιθέμενη αξία του. Και θα πρέπει τα επόμενα έτη να το κάνετε αυτό και σας παρακαλώ να μου πείτε τι έχετε υπόψη σας να κάνετε. Και μια τελευταία ερώτηση. Είστε έτοιμοι εσείς προσωπικά να σκεφτείτε κάποια μέτρα που να επιτρέπει στη δική μας Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγή. Ευχαριστώ. Ξεκινάω με το τελευταίο ερώτημα. Βεβαίως ε, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχυνθεί η διαδικασία απαλλαγή. Ε, και έχω συζητήσει με το θέμα αυτό επανειλημμένα με την κυρία Χολμάια ε, κοιτάξτε, το δικό μας το πρόβλημα είναι ότι δεν εξαρτάται όμως μόνο από εμάς τους δύο, δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο από το Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο σημαντικότερος εταίρος ε, σε αυτή τη σχέση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αυτήν ελέγχουμε. Και ε, είμαστε ανεξάρτητοι από τους αριθμούς που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι αριθμοί, τα στοιχεία έρχονται αρκετά καθυστερημένα. Ε, ίσως ε, θα έπρεπε ε, κατά διάρκεια αυτής της θητείας να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία από κοινού δηλαδή, να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και επίτροπο για τον προϋπολογισμό και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε επιτάχυνση της διαδικασίας. Θέλω να πιστεύω θα υπάρξει και αλλαγή του financial regulation. Ε, πάντως εμείς το θέλουμε αυτό. Αλλά βέβαια σε τελική ανάλυση αυτό είναι απόφαση του νομοθέτη. Για το τελευταίο ερώτημα. Τώρα για το ερώτημα τι μπορεί κανείς να βελτιώσει. Έχω ένα κλασικό παράδειγμα. Όταν το 2014 εξελέγει για πρώτη φορά στο συνέδριο, τότε τέλη Απριλίου θεσπίσαμε μία έκθεση η οποία εμφανίστηκε σε μία συνέντευξη τύπου και αφορούσε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ε, δύο εβδομάδες νωρίτερα είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών. Είχαμε λοιπόν την ε, απόφαση η οποία είχε δρομολογήσει αυτή την ε, τραπεζική ένωση. Λάθος όμως η χρονική στιγμή. Αυτό ήταν λάθος και γι' αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό να μην επαναληφθεί. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια αυτό που κρίναμε ότι είναι πολύ σημαντικό είναι ο χρονισμός, το timing. Δηλαδή να εμφανίζονται εκθέσεις όταν το περιεχόμενό τους έχει νόημα και όχι απλά να αναφερόμαστε και να διαφωτίζουμε σε κάτι που αφορά στο παρελθόν, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας επιδιώκουν καλύτερους νόμους. Για το μέσο άνθρωπο. Αναφέρθηκα ήδη στην εισαγωγή μου και επίσης ε, και απαντώντας σε ερωτήσεις. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας προς τα έξω και το έχουμε ήδη επιτύχει. Έχουμε ε, προτάσεις, ε, σας είπα και από το peer review περιμένουμε και άλλες, αλλά όμως υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο θεμελιώδης πρόβλημα είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο μικρότερος από τους 7 θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίπου 900, πάνω από 900 εργαζόμενους. Δύο-τρει ασχολούνται με τον τύπο. Καλή δουλειά τους. Όμως αυτοί υπηρετούν 28 διαφορετικά ε, τοπία και μέσα ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 28, δηλαδή διαφορετικά κράτη-μέλη. Γιατί είναι ξεχωριστά όλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος έχουν ένα ή περισσότερα γραφεία με τα οποία ε, ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωση. Όμως ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είμαστε πολύ μικρός ο οργανισμός. Ως εκ τούτου οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Πάντως προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε ε, μια πόλη, το Λουξεμβούργο, πολύ καλοί, οργανωμένοι, εκεί βρισκόμαστε, όμως είμαστε αποκομμένοι από τα μέσα ενημέρωσης, ε, που είναι εδώ. Εδώ στις Βρυξέλλες είναι όλοι οι ανταποκριτές των μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Εδώ γίνονται οι εκθέσεις, ε, από εδώ γίνονται οι αναφορές, άρα δηλαδή αναγκαστικά υπάρχει αυτό, αυτή η απομόνωση. Εμείς βέβαια προσκαλούμε δημοσιογράφους ε, που έρχονται και μας επισκέπτονται και άλλους θεσμούς. Πολλά κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά σας λέω ότι υπάρχει αυτό το εγγενές μειονέκτημα στη δική μας την περίπτωση. Και μπορείτε επίσης και να δείτε στην ε, έκθεσή μας των δραστηριοτήτων ότι έχουμε επεκταθεί πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 50% της ενημέρωσης γίνεται πλέον μέσω αυτών και ως εκ τούτου έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, αλλά βέβαια οι δυνατότητες του ελεγκτικού συνεδρίου για τα μέσα κοινωνική δικτύωσης δεν είναι ατελείωτες. Ε, Εμεί δεν μπορούμε να γράφουμε στο Twitter αυτά που γράφουν άλλοι, απλά. Ως εκ τούτου και εκεί υπάρχουν περιορισμοί για μας ε, για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ζούμε με αυτά τα handicap, με αυτά τα εμπόδια και προσπαθούμε, έχοντας αυτά κατά νου, να επιτύχουμε το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Πέξα έχει το λόγο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μαζί σας. Ε, θα ήθελα να συνταχθώ με τους ε, προλαλήσαντες συναδέλφους και να τονίσω πως άκουσα με μεγάλη χαρά πως όλο και περισσότερες γυναίκες ε, παίρνουν όλο και καλύτερες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ελπίζω πως ε, αυτό το 21-7 που είναι η σημερινή κατάσταση στο μέλλον θα αναστραφεί έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Έχω μια ερώτηση ή μάλλον καλύτερα να μου σχολιάσετε εσείς ένα στατιστικό στοιχείο ε, ενός πολιτικού θέματος επίτροπο για ε, προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή έχουμε Γερμανό ε, από το ΕΛΚ. Ε, Επιτροπής προϋπολογισμών, έχουν προϋπολογισμών Γερμανία CSU. Ελεγκτικό συνέδριο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτες και αυτός και στην επόμενη ε, θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από το Λαϊκό Κόμμα Αυστριακός για τον προϋπολογισμό. Πώς σας φαίνεται που είναι όλοι από την ίδια πολιτική οικογένεια και μάλιστα κάποιοι από το ίδιο ε, κράτος. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ο ένας τον άλλο. Προφανώς και μπορούμε. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ξέρετε, ο πιο αυστηρός επικριτής της κυρίας Φόντερ Λάιν στη Γερμανία είναι το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο και πρόεδρος ε, είναι ο πρώην ε, εκπρόσωπος του Τσεντεού Τσεσού στο ε, Γερμανικό Κοινοβούλιο. Άρα δηλαδή βλέπετε ε, τα πράγματα νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφή. Εγώ το 2014 όταν εξελέγη στο ελεγκτικό συνέδριο, δύο μήνες πριν από την εκλογή μου, εγκατέλειψα όλες μου, όλα μου τα αξιώματα στο κόμμα και δεν ασχολήθηκα πλέον με αυτά. Άρα δηλαδή είναι αυτονόητο. Όταν λαμβάνει κανείς ένα τέτοιο καθήκον, προφανώς και πρέπει να είναι αμερόληπτος, ουδέτερος πολιτικά, έτσι πρέπει να ζει. Ε, την κυρία Λάιν την γνώρισα πριν από δύο εβδομάδες. Τότε την πρώτο είδα. Δεν την είχα ξαναδεί. Γιατί η κυρία Λάιν ασχολιόταν στο κόμμα με τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που ασχολιόμουν εγώ, από άλλη, άλλο κρατήδιο, Τίποτα, καμία σχέση, καμία επαφή. Ε, και νομίζω αυτή είναι και η άποψη των ε, συναντέλφων μου ότι δεν με επιβαρύνει καθόλου η σχέση με την κυρία Φοντελάν. Γιατί αν με επιβάρυνε, ε, ξέρετε, νομίζω ότι δεν θα με είχαν εκλέξει με τόσο μεγάλη πλειοψηφία πριν από λίγο καιρό στη θέση του Προέδρου του Ελληνικού Συνεδρίου. Καμία σχέση λοιπόν. Δεν νιώθω καμία επιβάρυνση από την κυρία Φοντελάν. Και θέλω να πω ότι και η κυρία Γκρέσλε και αυτή ήταν Γερμανίδα ο κύριος Χαν, λάθος το είπατε εκεί, δεν είναι Γερμανός, είναι Αυστριακός και μόνον αυτό, αλλά το θεωρεί και πολύ σημαντικό ε, που είναι Αυστριακός. Έτσι λοιπόν κάπως βελτιώνει την κατάσταση, δεν έχουμε μόνο Γερμανούς, έχουμε και Αυστριακούς. Πολύ ωραία. Να ερωτήσω αν έχετε να υποβάλλετε άλλες ερωτήσει Ο κύριος Αντινόλφη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω, εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα οποία μας είπε ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, την εμπειρία του και την ηλικία του, γιατί όταν ε, έχει κανείς και αυτή την ηλικία προφανώς και έχει και μεγαλύτερη εμπειρία. Ε, παρατηρώ με ικανοποίηση ότι η Γερμανία εκπροσωπείται μια χαρά ε, στο ελεγκτικό συνέδριο, με την κυρία Φοντελάνη στην Επιτροπή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, η εκπροσώπηση είναι πάρα πολύ ουσιαστική όσον αφορά τουλάχιστον τη Γερμανία. Από αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου κατέστησε σαφές ότι έχουμε θεσμούς όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασκείται κάποια κριτική έναντι αυτού, δηλαδή ότι κατά κάποιον τρόπο ε, δεν ε, κοινοποιείται, δεν γίνεται ουσιαστική η παρουσίαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί τα μέσα ενημέρωση βρίσκονται εδώ στις Βρυξέλλες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο πράγματι είναι στο Λουξεμβούργο και πράγματι υπάρχει αυτή η κριτική πολιτική που ασκείται έναντι όλων των υπόλοιπων ε, κοινοβουλίων, εγώ θα ήθελα να μας πείτε ποια ακριβώς ε, είναι η άποψή σας. Προ αποφυγή παρεξηγήσεων. Εγώ δεν είπα να φύγει από το Λουξεμβούργο το ελεγκτικό συνέδριο, διότι μα αρέσει πάρα πολύ εκεί και δεν θέλουμε καθόλου να φύγουμε. Και δεν είναι τυχαίο ε, που ε, κάποιοι θεσμοί, ε, όπως το ελεκτικό συνέδριο ή το δικαστήριο, που πρέπει να είναι εκτός της καθημερινής πολιτικής σκηνής ε, και <laughs> τους προστατεύουν λίγο και τους βάζουν σε άλλες πόλεις. Αυτό έχει το μειονέκτημα όμως για μας, ότι δεν έχουμε πρόσβαση στους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι εκεί που συμβαίνουν τα γεγονότα. Ε, δυστυχώς με αυτό το μειονέκτημα θα πρέπει να ζήσουμε. Και αυτό όμως εξηγεί το λόγο για τον οποίο υπάρχει καμιά φορά δυσκολία ε, ε, στο να αντιλαμβάνεται ο μέσο Ευρωπαίος πολίτης και να γνωρίζει τι είναι το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο καλό να πάτε, είστε ελεύθερο. Okay. Draußen wartete schon der... Περιμένει έξω ο ο επόμενο υποψήφιος, ο κύριος Μιλιώνη. Welcome to the committee. Καλωσορίσατε ορίσατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, στην ακρόασή σα. Είστε ο ε, Έλληνας υποψήφιος. Ο εισηγητή σα είναι ο κύριο Σάντρο Ρονάη από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. You have the floor. Παρακαλώ κύριε Μιλιάνη, έχετε το λόγο. Um, thank you. Madam Chair. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή η ευκαιρία που έχω να σας ομιλώ ως υποψήφιος για το διορισμό μου ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Τελευταία εξαετία έκανα ό,τι μπορούσα για να ανταπεξέλθω στις υψηλές προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών και να σφυριλατήσω στενή σχέση με τους εκπροσώπους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Is... Πιστεύω ακράδαντα ότι ε, μπορούμε να βοηθήσουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη σωστή κατεύθυνση. Σωστά, η συνθήκη ζητάει από τους ελεγκτές να είναι ε, ανεξάρτητοι επαγγελματίες με υψηλά προσόντα και με αδιαμφισβήτητη ανεξαρτησία. Από μία 20 και πλέον ε, ήμουν δικαστής στο Ελληνικό Ελεκτικό Συνέδριο πριν γίνω αντιπρόεδρος. Ως δικαστής έχω ισχυρή ανεξαρτησία και στο θεσμικό μας πλαίσιο αυτό είναι παράδοση ε, ε, εκτός από την καριέρα μου αυτή, ε, δίδαξα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών οικονομικό δίκαιο και έχω κάνει και διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα για τη δημόσια διοίκηση και τον οικονομικό έλεγχο. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όταν με διορίσατε μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου πριν από έξι χρόνια που ήρθε σε μια περίοδο κλειδί ε, αυτό για μας. Ε, βάλαμε τον Ευρωπαίο πολίτη στην καρδιά της στρατηγικής μας, επιλέξαμε θέματα που είναι ε, πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων και ενισχύσαμε την παρουσία μας στα παραδοσιακά μέσα αλλά και στα κοινωνικά μέσα. Στο πρώτο τμήμα όπου προεδρεύω αυτή τη στιγμή, έχει διευρύνει τις αρμοδιότητές του ε, ε, πέρα από τις αρχικές που ήταν η κοινή γεωργική πολιτική, καλύπτουμε και ευρύτερα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Ως εισηγητής για τους φυσικούς πόρου στην ετήσια έκθεση εργάστηκα για να πιάνει περισσότερο τόπο ο έλεγχος που κάνουμε. Ε, την τελευταία τριετία καταφέραμε να δώσουμε ε, θετική δήλωση αξιοπιστία για τις άμεσες ενισχύσεις, αλλά ε, είπαμε ότι υπάρχουν και τομείς υψηλού κινδύνου και τους φωτίσαμε. Ε, απελευθερώσαμε ε, πόρους από την συμμόρφωση για να προχωρήσουμε προς την απόδοση. Ε, διασταυρωμένη συμμόρφωση, ε, θέματα υποδομών ε, και άλλα θέματα γεωργικής πολιτικής ήταν αυτά που συγκέντρωσαν την προσοχή μας. Εκτός αυτού και το περιβάλλον που κάναμε λογιστικό έλεγχο ε, για την βιολογική γεωργία, για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τις περιοχές Natura 2000. Καθώς επίσης και μια έκθεση για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που επίκειται η δημοσίευση της. Αυτές οι εκθέσεις οδήγησαν στην καλύτερη διαχείριση των πολιτικών και των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κατά την πάροδο αυτών των ετών, με χαρά είδα να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο οι εμπλεκόμενοι ε, για τις εκθέσεις μας, όχι μόνο από τη δική σας επιτροπή, αλλά και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο τύπος, ε, η κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα ε, όταν ήταν θέματα που τους αφορούσαν άμεσα. Αυτό τι δείχνει, ότι αυξάνεται η σημασία μας και τελικά ο θετικός αντίκτυπος που έχουμε στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Για να έχει νόημα η παρουσία μας θα πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Ακόμα ανακάμπτει η οικονομία από την κρίση που ξέσπασε το 2008. Τα θεσμικά μας όργανα, τα ευρωπαϊκά ή ακόμα και οι εθνικοί θεσμοί ε, καλούνται να βρουν λύσεις. Ε, τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρομέτρου είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι ανακάμπτει η εμπιστοσύνη στο δικό μας θεσμικό όργανο. Έχουμε όμως ακόμα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Εκτός από τα οικονομικά προβλήματα και τα κοινωνικά, οι πολίτες μας ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη, για την ε, ε, επιδείνωση του περιβάλλοντος και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία τους. Με άλλα λόγια, οι πολίτες ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των σημερινών ε, δημοσίων πολιτικών. Και πιστεύω ότι οι νομοθέτες, η εκτελεστική εξουσία και οι ελεγκτές, ο καθένας από τη σκοπιά του και βάσει της εντολής του, θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο πιο σημαντικό για την εμπιστοσύνη των πολιτών με ανεξαρτησία, με επαγγελματισμό, θα ελέγχουμε εμείς τα οικονομικά και αυτό μπορεί να ε, βεβαιώνει καλύτερα και να καθησυχάζει τον πολίτη για το τι γίνεται και τι απομένει να γίνει. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σάντορ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο και μια και έχω αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να καλωσορίσω εκ μέρους των σοσιαλιστών ε, τον κύριο Μιλιών. Είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε το θέμα ε, εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Είχαμε και την προηγούμενη παρουσίαση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως εσείς έχετε τις ε, γνώσεις και την εμπειρία που είναι απαραίτητες για να ε, καλύψετε αυτή τη θέση. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει τα τελευταία έξι χρόνια το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών έχουμε το καθήκον να παρακολουθούμε έτσι ώστε οι δαπάνες και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δίδονται με διάφορο τρόπο και ε, υπέρ των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερέντων. Χαίρομαι που η προτεραιότητά σας είναι καλή σχέση μαζί μας και περισσότερο βαθιά ε, σχέση στο μέλλον, αλλά έχω και μία σειρά από ερωτήσεις που θα ήθελα να σας κάνω σχετικά. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εσείς λέτε πως ε, καθυστερούν πολύ οι εκθέσεις αναλύεται τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και βρίσκεται ότι πολλές φορές υπάρχουν κενά. Δεν νομίζετε πως πολλές φορές έχουμε επικάλυψη εργασιών σε πολλούς χώρους. Υπάρχει κάποια λύση ε, στο μυαλό σας γι' αυτό, ώστε να μην έχουμε επικάλυψη, έτσι ώστε να μην έχουμε επανάληψη ε, ελέγχων που έχουν γίνει αφενός, γνωρίζοντας πώς θέλουμε να μειώσουμε το διοικητικό βάρος. Τι εργαλεία έχουμε που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των επικαλύψεων. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Εσείς ήσασταν πρόεδρος τμήματος ε, για την προηγούμενη κοινή γεωργική πολιτική, την ΚΑΠ. Στην επόμενη ΚΑΠ θα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ε, με ποια εργαλεία θα πετυχαίνουν τους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη. Σήμερα στους New York Times λέει πως μια σειρά κρατών από την Ανατολική Ευρώπη ή οι κυβερνήσει του και οι ολιγάρχες που συνδέονται με τις κυβερνήσεις κάνουν απατηλή χρήση των ευρωπαϊκών ε, κονδυλίων ε, για κερδοσκοπικούς λόγους και λάπτοντα τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πώς το ευρωπαϊκό χρήμα θα χρησιμοποιείται με τους στόχους που έχουμε θεσπίσει, γνωρίζοντα τα όσα γίνονται. Ποια είναι η μεθοδολογία την οποία θα προτείνετε έτσι ώστε να προετοιμαστούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και έχω και μια τρίτη τελευταία ερώτηση. Θεωρείτε πω είναι σημαντικό να συνεργάζεστε με τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια έτσι ώστε τα εθνικά ελεκτικά συνέδρια να μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στο ευρωπαϊκό. Συνεργασία, για παράδειγμα, για τη μείωση ε, των ε, εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου, στόχοι του 2030, τάσεις οι οποίες εμφανίζονται στα κράτη-μέλη και τα οποία θα πρέπει να, και οι οποίες θα πρέπει να σας γνωστοποιηθούν. Εφαρμογή των κρατών μελών, των στόχων που έχουμε για την κλιματική αλλαγή. Αυτές ήταν οι ερωτήσει μου και θα ακούσω με χαρά τις απαντήσεις σας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Μιλιώνη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, σχετικά με την καθυστέρηση των εκθέσεων ε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ε, εμείς σε ό,τι αφορά την, ε, την, την ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλουμε κάθε χρόνο σε εσά, έχουμε βελτιώσει το χρόνο από τον Νοέμβριο το, την υποβάλλουμε τον Οκτώβριο. Αυτό βέβαια ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα αλλά θα μπορούσε αυτό να γίνει καλύτερο, να περάσουμε σε καλύτερους χρόνους εάν εκμεταλλευόμασταν τα ε, control systems των κρατών μελών. Η δικιά μας δουλειά ε, στηρίζεται στην, ε, στα control systems των κρατών μελών. Αν αυτά βελτιωθούν, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση, βέβαια και από την Κομισιόν, να έχουμε γρηγορότερα την πληροφορία την οποία ζητάμε. σε ό,τι αφορά, αφορά τώρα τις αυτό ήταν για την ετήσια έκθεση. Ό,τι αφορά τις ειδικέ εκθέσεις, ε, το ζήτημα είναι πως εκεί έχουμε ένα όριο από τον δημοσιονομικό κανονισμό των 13 μηνών. Αυτό, αυτόν προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε. Δεν τον έχουμε πλησιάσει ακόμη σε όλες σε όλο το φάσμα των ε, εργασιών στο performance που κάνουμε. Ε, είμαστε το 18, είχαμε πλησιάσει τους μέσο όρο το, 15,2 μήνες, αλλά προσπαθούμε όλο περισσότερο να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο. Σε ό,τι αφορά το, την επικάλυψη των εργασιών, πραγματικά εμείς παρατηρούμε πως υπάρχει επικάλυψη των εργασιών σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ε, ε, εθνικών ελέγχων, αλλά και των ελέγχων που κάνει η Επιτροπή. Σε αυτό το, εκεί στο στο οποίο προσπαθούμε να συμβάλλουμε περισσότερο είναι να αναπτύξουμε τον single audit ή το attestation approach, όπως λέμε, δηλαδή να στηριζόμαστε στην ελεγκτική εργασία την οποία κάνουν άλλοι ελεγκτικοί φορείς ή της Κομισιόν ή των εθνικών ε, των κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη στην κοινή αγροτική πολιτική έχουμε το, το, πρώτο level είναι οι paying agencies, το δεύτερο level είναι certification bodies. Τα certification bodies αυτά δίνουν ε, από, το, από, το 95 και, από 2015 και μετά υποχρεωμένα να δίνουν μια opinion στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη, το legality και regularity. Αυτό θα ήταν μεγάλο επιτεύγμα εάν ακολουθούσαν, αν η πληροφορία που έδιναν ήταν reliable. Μέχρι τώρα δεν είμαστε τόσο, δεν είμαστε τόσο ικανοποιημένοι στην αγροτική πολιτική από τα certification bodies. Στο cohesion γίνεται από το, 2017, από το γίνεται, ε, ε, στηρίζονται στην δουλειά των, ε, των ε, εσωτερικών ελεγκτών των ελεγκτών, εννοώ που γίνεται, που είναι, όχι των εσωτερικών ελεγκτών, των ελεγκτών των κρατών μελών, των, ε, των οποίων που δίνουν τα κράτη-μέλη και εκεί έχει προχωρήσει η δουλειά. Σε ό,τι αφορά την ε, κοινή γεωρική πολιτική υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια με 30 transactions από το, από το 2019 να πετύχουμε αυτό το είδο, να στηριζόμαστε δηλαδή στη δουλειά των άλλων και να μην έχουμε αυτή την επικάλυψη. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΚΑΠ, η ΚΑΠ πραγματικά τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει με το καινούριο, με, την, με, το, με το καινούριο delivery model του ΚΑΠ, της ΚΑΠ μετά το 2020 να, να, να, να καταθέτουν strategic plans. Η Κομισιόν, το πρόβλημα είναι πως η Κομισιόν δεν έχει ακόμη ε, υπάρχουν, υπάρχει μια έλλειψη καθαρότητα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα της Κομισιόν να ελέγχει αυτά τα strategic plans για να μπορούν να, να ελέγχονται από το, σε κεντρικότερο επίπεδο. Τώρα για το ζήτημα πραγματικά που ε, θέτεται για, το, για, τα, για κάποια ζητήματα που έχουν ανακύψει στην Ανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αρπαγή κάποιων ε, εκτάσεων, δημοσίων εκτάσεων και την πώληση σε, ε, σε ιδιώτες και ούτως ώστε αυτοί οι ιδιώτες να επωφελούνται από, την, ε, από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Αυτό θα μπορούσε να, να είναι ζήτημα βέβαια του κοινοτικού, του ευρωπαϊκού νομοθέτη να τα ρυθμίσει. Εμείς όταν βρίσκουμε ζητήματα fraud τα παραπέμπουμε κατευθείαν στην ΟΛΑΦ ε, και η ΟΛΑΦ συνεχίζει την, την, την, ε, τις εργασίες της. Ε, αλλά πολλά από τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα κυρίως της εσωτερικής ε, τάξεως των κρατών μελών. Το, το, το δικαστικό σύστημα κάθε κράτους μέλους επιλαμβάνεται. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία με τα ε, εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, αυτό είναι ένα μεγάλο long-term vision για το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο συνεργάζεται σε επίπεδο Eurozai με τα, ελεγκτικά, με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. υπάρχουν ε, liaison officers οι οποίοι, έχουν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρουν στα κράτη-μέλη, στα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια την πληροφορία από, τα, από, τα, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την υποβολή, υποβολή προδικαστικού τρόπων την ερωτήματο, όπω συμβαίνει με τα δικαστήρια που υποβάλλουν προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί ε, Νομίζω πως είναι πολύ τολμηρό, πολλοί το έχουν σκεφτεί αυτό, αλλά δεδομένου ότι το ε, ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δικαστικές αρμοδιότητες. Πολλά από τα ελεγκτικά εθνικά συνέδρια, αρκετά, κυρίως του Νότου, έχουν δικαστικές αρμοδιότητες. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να συνδυαστεί αυτό το ζήτημα. Α, αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στον Τόμας Στεχόφσκι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλιώνη. Ήταν μία απάντηση η οποία απάντησα στα θέματά μας. Στα ερωτήματα που απαντήσατε μιλάτε για την εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη για μας είναι κομβική. Εμείς πήγαμε πολλές αποστολές στην Ελλάδα και είδαμε πολλά πολλά σφάλματα και λάθη. Ήσασταν το μέλος της Εθνικής ε, Αρχής Ελέγχου για πάρα πολλά χρόνια. Είστε πάρα πολύ έμπειρος. Έχετε πολλές δημοσιεύσεις, βιβλία. Ερωτώ λοιπόν το εξής. Εμείς πήγαμε σε αποστολή για το Μετρό της Θεσσαλονίκης και ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί, ακόμα έχει προβλήματα, έχουμε ακούσει όλες τις εξηγήσει. Τι πιστεύετε, ποιο είναι το σημείο κλειδί στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για ποιο λόγο δεν είμαστε τόσο πετυχημένοι, γιατί δεν έχουμε επιτυχίες σε πολλά από αυτά τα project τα οποία έχουμε χρηματοδοτήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς θα προωθήσετε εσείς ε, στο ελληνικό κοινό την ιδέα πως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάνουν άριστη δουλειά και θέλουν να αλλάξουν πολλές από αυτές τις ε, αδυναμίες Γιατί είναι ακόμα στα σκαριά και δεν έχουν τελειώσει ε, με τον ικανοποιητικό τρόπο. Επίσης, δεύτερη ερώτηση. Γιατί θέλετε να είστε άλλα έξι χρόνια στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάνατε ε, εξαιρετική δουλειά. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Και ίσως λίγο προκλητική η επόμενη ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσετε εσείς πράγματι ότι θέλετε να μείνετε και κάτι θέλετε να κάνετε. Όχι ότι θέλετε να μείνετε μόνο για τα επόμενα έξι χρόνια επειδή είναι η τέλεια δουλειά. Επίσης, θέλω να δω και τις σύγχρονες ελεγκτικές μεθόδους. Ξέρω πως έχετε εμπειρία και έχω διαβάσει ένα από τα άρθρα σας και μιλάτε ε, για κάθε τα θέματα επίσης, όχι μόνο οριζόντια και ε, τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Οπότε εσείς αυτό πώς θα το αλλάξετε, προς ποια κατεύθυνση, γιατί πολλές φορές έχετε επικρίνει το γεγονός πως έχουμε εξαιρετικά αεροδρόμια, στα οποία όμως δεν πετάνε αεροπλάνα. Οπότε, ε, για ποιο λόγο είναι εκεί. Λιμάνια στην Ισπανία, αλλά τα καράβια πάνε στα λιμάνια τα μαροκινά αντί στα ισπανικά. Ε, αυτά είχα ως συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα περιμένω τις απαντήσεις σας. Thank you. Ε, ε, ε, φυσικά η, το τράστ, η εμπιστοσύνη είναι κομβική για την πρώτον και κύριο να εμπιστεύεσαι αυτόν στον οποίο στέλνεις τα χρήματά σου πως ε, τα χρήματα αυτά θα, δεν θα γίνουν μόνο με νόμιμο και ε, κανονικό τρόπο, αλλά και με τον πλέον αποδοτικό τρόπο θα χρησιμοποιηθούν. Ε, στην Ελλάδα το πρόβλημα α, ως μέλος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου εμείς είχαμε πολλές φορές και πριν την κρίση επισημάνει ζητήματα σε εκθέσεις μας αλλά δεν βρίσκαμε από την άλλη πλευρά ευήκονους, ευήκονους ε, Ίσως στη χώρα μου υπάρχει ένα πρόβλημα ε, λειτουργίας των θεσμών, αλλά δεν μπορώ τώρα να εκταθώ εδώ σε πράγματα ε, που αφορούν την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά βέβαια την Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη έχει το πρόβλημα πως, ε, που έχει όλος ο Νότος, πως είναι τα διάφορα layers της ιστορίας. Είναι η αρχαία πόλη, η ρωμαϊκή πόλη, η βυζαντινή πόλη. Όταν έσκαψαν βρήκαν διάφορα πράγματα. Μετά η κάθε κυβέρνηση είχε την, το δικό της ε, πλάνο σχετικά με την πώς θα αξιοποιηθούν αυτά, αυτές οι αρχαιότητες. Ε, όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα με ένα άλλο αδύρυτο, το δυσκολότερο πρόβλημα που είναι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα δημιούργησαν αυτές τις καθυστερήσεις. Ας ελπίσουμε πως τώρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ε, ε, τι κάνουμε βέβαια για να γίνει το ελεγκτικό, η δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου πιο γνωστή στο ελληνικό κοινό. Ε, προσωπικά εγώ άρχισα τις ε, ε, παρουσιάσεις των ε, προϊόντων μας που λέμε, των, των εκθέσεων που κάνουμε, των opinions που δίνουμε, των ειδικών εκθέσεων που δημοσιεύουμε ε, στη Βουλή. Ε, η Βουλή μέχρι τώρα, μέχρι πριν από μένα, δεν δεχόταν να, να, να ακούσει. Ε, νομίζω πως αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Παρουσιάζω στο Πανεπιστήμιο ε, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ε, τις εκθέσεις και όχι μόνο τις εκθέσεις αλλά και, με, και τη μεθοδολογία την οποία ε, ε, αναπτύσσουμε κατά, την, ε, κατά τον έλεγχο που κάνουμε. Και αυτό είναι περισσότερο και είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο άρχισε κυρίως από τον συνάδελφό μου, τον, Μπρένικ, τον κύριο Μπρένικ Μάγερ, πως να θέσουμε στο, στο, στο δικαιικό σύστημα μια άλλη πτυχή, τον έλεγχο ως ένα τέταρτο ε, πυλώνα ε, εκτός από την νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική εξουσία, να, να πούμε και πως υπάρχει και η ελεγκτική εξουσία σαν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω αυτό ε, έγινε γνωστό και στο, ε, τουλάχιστον στο, στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στο χώρο του, του Κοινοβουλίου. Γιατί θέλω άλλα έξι χρόνια. Γιατί νομίζω πως αρχίσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα στο πρώτο τμήμα στο οποίο είμαι, με πρωτοβουλία του συναδέλφου μου, του Φιλβινόουεν, που όταν άρχισε με το πρώτο landscape review ε, για το energy και, και, και, το, και το climate change άνοιξε για το πρώτο τμήμα ένας καινούριο ορίζοντας και έκτοτε έχουμε βάλει στην ατζέντα μας για τις πλημμύρες, έχουμε βάλει για το, ε, το, και την ερημοποίηση, ε, εγώ έχω κάνει για το greenhouse gas emissions και προχωρούμε. Νομίζω πως αυτό είναι ένα καλό, μια, ένα καλό, μια καλή πορεία που πρέπει να συνεχίσουμε για τις, modern, ε, ε, για τις ε, μοντέρνες τεχνικές ελέγχου. Οι μοντέρνες τεχνικές ελέγχου είναι ένα μεγάλο challenge για το ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς χρησιμοποιούμε πολύ το, διάφορα το satellite images, χρησιμοποιούμε όρθο κυρίως στην, στην αγροτική πολιτική με το LPIS, ε, έχουμε μειώσει με, όλα αυτά, με όλους αυτές τις μοντέρνες τεχνικές τους ε, on the spot ε, ελέγχους που σημαίνει κάνουμε μεγάλο, μεγάλο saving στα resources μας. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας όλες αυτές τις μοντέρνες τεχνικές έχουμε, έχουμε φτάσει στο μισό από τους ε, on-the-spot ελέγχους. Ε, ένα άλλο πράγμα για να γίνει πιο μοντέρνος ο έλεγχος είναι παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε το Sentinel Images που βέβαια δεν είναι εμείς υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, είναι η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό το παρακολουθούμε στην αγροτική πολιτική που είμαι ε, αυτά τα χρόνια υπεύθυνο. παρακολουθούμε τα, τα, τα, τα, τι achievements έχουν επιτευχθεί είναι για το ζήτημα του αεροδρομίου, για το ζήτημα ε, των, λιμανιών. Είναι δυστυχώς δύο περιπτώσεις, οι πιο, οι πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις που ε, διαπιστώσαμε με εκθέσεις μας, ε, όχι στο δικό μου τμήμα, αλλά στο δεύτερο τμήμα, πως ε, οι objectives δεν ήταν ε, σωστοί, οι indicators δεν ήταν σωστοί, και έγιναν πράγματα τα οποία μάλιστα στην Ελλάδα υπάρχουν σε απόσταση ξέρω εγώ, 50 χιλιόμετρων δύο αεροδρόμια. Ε, αυτό είναι καλό βέβαια για, για τους δημάρχους αλλά όχι για, τις, ε, για την ανάπτυξη και την, ε, ε, των πολιτικών μας. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Λιβιέ Σαστέλ. Όχι, ο κύριος Μποαγιέ πρώτος. Ε, κυρία Πρόεδρε, δεν με θέλετε καθόλου από το πρωί. Ε, θα μιλήσω όμως. Πάντα σε κάποιον άλλον θα δώσετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Μιλιώνη και για τις γραπτές και για τις προφορικές σας απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ κατατοπιστικές. Άκουσα ότι ενδιαφέρεστε πολύ για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τα γεωργικά ζητήματα, τα οποία είναι αλληλένδετα με τα προηγούμενα και όλοι πιστεύουμε ότι αυτά τα θέματα θα κυριαρχήσουν στην κοινοβουλευτική περίοδο που τώρα αρχίζει. Έχω μια απλή ερώτηση να σας κάνω. Για αυτά τα θέματα περιμένουν οι πολίτες από εμά και από εσά να δείξουμε αποτελεσματικότητα και διαφάνεια για τα θέματα αυτά και για πολλά άλλα. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω το εξής. Τι χρειάζεστε ή τι θα μπορούσατε να περιμένετε από εμάς, τους νομοθέτες, για να σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε καλύτερα σε αυτή την αποστολή και σε αυτούς τους στόχους, ιδιαίτερα τους περιβαλλοντικούς και γεωργικούς. Ευχαριστώ. Τι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον νομοθέτη. Πρώτον και κύριον να είναι το simplification. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, διότι στην αγροτική πολιτική έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους της υπαίθρου, από εκεί προέρχομαι και το ξέρω, ε, που θα πρέπει τους ανθρώπους να τους δίνουμε την πληροφορία με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Ε, καταλαβαίνω πως τα διάφορα layers νομοθετήσεως δημιουργούν προβλήματα, αλλά νομίζω πως είναι ζήτημα που αφορά εσάς και αφορά και το Κονσέι για να γίνει το πράγμα πιο απλό. Ε, αυτό θα έλεγα πως είναι και βέβαια, και βέβαια χρήματα. Ας πούμε στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής ε, στο Climate Action ε, υπάρχει ένα παράπονο πως είναι λίγα τα χρήματα που δίνονται. Είναι λίγα τα χρήματα. Ε, δεν, ε, βέβαια, ε, δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό, αλλά βλέπει κανείς πως υπάρχουν... Η κοινή αγροτική πολιτική έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, Βλέπει ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν ειδικού τομεί θα πρέπει ίσως να ενισχυθούν. Αυτά θα μπορούσα να απαντήσω. Vielen ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα τίθεται το ερώτημα αν ο κύριος Πέκτσα θέλει να κάνει ερώτηση, βεβαίως. Good morning and thank Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα τον καινούριο σας ρόλο. Να σας πω πως εκτίμησα ιδιαίτερα την η υποψηφιότητά σας γιατί δεν έχετε πολιτική ε, σχέση με τρέχοντα κόμματα και έτσι μπορούμε ε, να εξασφαλίσουμε την αμεροληψία. Επίσης, μου αρέσουν οι επαγγελματίε όταν ελέγχουν τα δημόσια ή οικονομικά. Τις αρχικές μου ερωτήσεις τις έκαναν κυρίως οι συνάδελφοι και τις έχετε απαντήσει. Μιλήσατε για τα προβλήματα τα οποία οδήγησαν ε, κατόπιν στην ε, ελληνική κρίση με τα δημόσια οικονομικά και αν κατάλαβα καλά δεν έχετε εισακουστεί από τις ε, ελληνικές αρχές. Πείτε μου, ποιοι θεωρείτε πώς ήταν υπεύθυνοι για το γεγονός ότι τότε αγνοήθηκαν οι εκθέσεις σας ή οι συστάσεις σας. σε ομολογώ. Ε, βέβαια, ε, κάναμε για σειρά ετών για σειρά ετών έχουμε μια ειδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων στο Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ε, τόσο είναι ένα είδος δήλωσης αξιοπιστίας, όπως λέγεται, όπως μια αντίστοιχη ορολογία, αλλά όχι ίδια, το ίδιο περιεχόμενο, και η ετήσια έκθεση. Ε, φοβούμε πως ε, δεν υπήρχε μια κουλτούρα να εισακούγονται όχι μόνο οι ελεγκτές στην Ελλάδα, που και στην Ελλάδα εμείς είμαστε δικαστήριο. Δηλαδή, ο Νότος έχει εφοδιαστεί για λόγους άλλους που δεν είναι της τρέ... Ε, ε, δεν μπορώ να τα εξηγήσω τώρα εδώ, ε, είναι εφοδιασμένος με ελεγκτικά συνέδρια ως δικαστήρια. Υπάρχει λόγος για ποιο λόγο. γιατί. Παρά το γεγονός πως ήμασταν δικαστήριο, η εκτελεστική εξουσία δεν μας άκουγε. Ήταν ένα είδος έλλειψης κουλτούρας ελέγχου, θα έλεγα. Ε, το δε κοινοβούλιο πολύ αργά άρχισε να δέχεται... Ε, ήταν απλώς μια... Η αιτήσια έκθεση απλώς δινόταν στον πρόεδρο της Βουλής, χωρίς καμιά συζήτηση άργησε πολύ και με ανθρώπους που προήρχονται από εδώ, από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέβηκαν κατόπιν στην, στο Εθνικό Κοινοβούλιο και είχαν λόγο και μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν διατάξεις για να, οι... να εισακούγονται οι εκθέσεις του Ελληνικού ελληνικού Συνεδρίου. Ήταν μια έλλειψη κουλτούρας ελέγχου. Αυτό θα μπορούσα να πω, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Ω πρόεδρο θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση που ε, νομίζω ότι είναι σημαντική για την ανεξαρτησία των ε, δραστηριοτήτων σας στο ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει περίπτωση του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου που μας απασχολεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχαμε ασχοληθεί. Κατηγορούν τον κύριο αυτό της στατιστικής υπηρεσίας ε, πώς να το πω, ότι ήταν υπερβολικά ειλικρινής και τίμιος και έδωσε τα πραγματικά στοιχεία και όχι τα μαγειρεμένα που είχαν πιεστεί προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Και του καταμαρτυρούν και του προσάπτουν ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και στη Γερμανία καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και μάλιστα πρόσφατα η δική σας δραστηριότητα είναι ελεύθερη πιέσεων εκεί στο ελεκτικό συνέδριο ή ε, υφίσταστε κάποιες πιέσεις, γιατί μας ενδιαφέρει και για να σας προστατεύσουμε κιόλας, γιατί το, ε, τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να είναι ελεύθερα από κάθε πίεση έξωθεν, ακόμα και από το ίδιο το δικό τους κράτος μέλος. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να θέλει το κράτος μέλος να περιγράφονται διαφορετικά κάποια πράγματα όπως θα περιγράφει το ελεγκτικό συνέδριο. Θα καταλαβαίνετε αυτά τα θέματα, επιλαμβάνεται η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, και ανισχύει πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ερώτηση. Βέβαια είναι πάλι μια δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Ε, το ζήτημα είναι αν εμείς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είμαστε ε, ανεξάρτητοι από πιέσεις του εθνικού ή στο ελληνικό ελεγκτικό, στο εθνικό. Όχι. Για μένα τίθεται το ερώτημα εάν η ελληνική κυβέρνηση σας ασκεί πίεση για να αλλάξει ε, κάποιες εκθέσεις γιατί δεν της αρέσει ο τρόπος που τις γράφετε εσείς. Γιατί, ε, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην περίπτωση του κυρίου Γεωργίου και μένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανεξαρτησία ε, των μελών ε, του ελεγκτικού συνεδρίου ακόμα και είναι καινούργια κυβέρνηση. Ε, ε, η απάντησή μου είναι ούτε το διανοήθηκε ποτέ να το κάνει, ούτε το διανοείται, ούτε θα το διανοηθεί ποτέ, αλλά και αν το πράξει, ε, εγώ έχω, ε, έχω δείξει έχω, έχω, αποδείξει την ανεξαρτησία μου και στο ελληνικό και εδώ πως είμαι κουφός σε τέτοιου είδους. Το ζήτημα πιέσης. δεν, δεν υπήρξαν πιέσεις όμως ποτέ. Δεν υπήρξαν πιέσεις για να είμαι ειλικρινής. Σε ό,τι αφορά τον Γεωργίου είναι μια μακρά ιστορία η οποία εκθέτει ε, την χώρα. Ε, βέβαια τώρα η ελληνική διοίκηση λόγω των συνεχών αυτών διενέξεων, δικαστικών διενέξεων υποχρεώθηκε να, να του πληρώνει δικαστικά έξοδα όπως θα ξέρετε, ε, αυτό δείχνει κάτι. Τώρα, επί της ουσίας δεν μπορώ να λάβω. Αν και ο άνθρωπος συνέχεια, συνέχεια αθώνεται και στη συνέχεια η εισαγγελία του Αριοπάγου κάνει αναιρέσεις στο, στον Αριοπάγο και αρχίζει το πράγμα από την αρχή. Αλλά πλέον για να προστατευτεί ο άνθρωπος αυτός, ε, ίσως για την ειλικρίνειά του όπως είπατε, υποχρεώθηκε η ελληνική ε, διοίκηση να περάσει νόμο που να του πληρώνει όλα τα δικαστικά έξοδα. Αυτό είχα να απαντήσω. Καλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελοκληρώνεται εδώ η παρουσία ακρόαση και θα περάσουμε τώρα στη ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μιλιώνη. So, uh, Before we vote, I would uh, like to give the opportunity to... Πριν ψηφίσουμε, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία σε όλες τις πολιτικές ομάδες να κάνουν τις διαβουλεύσεις τους και να αποφασίσουν ότι θέλουν. Πέντε λεπτά φτάνουν ή χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Δέκα. Πέντε φτάνουν. Ωραία. Ρωτάω, δεν ξέρω. Πέντε λεπτά για τις ζυμώσεις των πολιτικών ομάδων.